So, ich glaube, wir können, wir können anfangen. Ich begrüße Sie, die zahlreichen Zuschauer. Σας καλωσορίζω. Είναι πολυπληθείς οι θεατές μεν, αλλά καλωσορίζω και τους ε, συναδέλφους στην κοινή επιτροπή μας, Επιτροπής Βιομηχανίας και ε, περιβάλλοντος, κοινή συνεδρίαση και έχουμε ένα κοινό μέλημα και καθήκον. Έκθεση πρωτοβουλίας θέλουμε να συντάξουμε και να περιγράψουμε πώς θέλουμε να είναι το μέλλον, να διαμορφώσουμε το πλαίσιο για την ενεργειακή και την κλιματική πολιτική. Έχει και νόημα αυτό. Για την υδρορογμάτωση ψηφίσαμε ε, το ίδιο ε, και ε, την ίδια μέρα μάλλον διαφορετικά πράγματα στις δύο επιτροπές, οπότε καλό είναι να συντονιζόμαστε και να έχουμε κοινέ θέσεις. Έχουμε τεράστια ευθύνη όλοι μαζί και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας, να βγαίνει κάτι κοινό με νόημα, να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και θα δείξει τι ε, επιτυχία θα έχουμε. Ελπίζω Έχω κάποιες ελπίδες και προσδοκίες ε, να αποθέσεις αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε και στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στην παρούσα να διαβάσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Έχουμε ορίσει και οι συγητές, δεν θέλω να μακρηγορώ εγώ. Θα δώσω το λόγο λέγοντάς σας ότι έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από εσθονικά και μαλτέζικα. Ε, χαίρομαι που βλέπω εδώ αριστερά την κυρία Σαρτόρη, συνάδελφο από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Ένα αλλάξει θα προεδρεύουμε, έτσι θα παίξουμε ε, την Προεδρία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην κυρία Σαρτόρη εισαγωγικά και μετά προχωρούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους βουλευτές. Και όπως θυμάστε και θυμήσατε πραγματικά κι εσείς στόχος της κοινή συνεδρίασης είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε οι συγιτές να μπουν σε αυτή την προσπάθεια της εκπόνησης της κοινή έκθεσης. Η Επιτροπή Ήτρα και Ένβη θα συνεργαστούν ε, σε αυτή την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της διαδικασίας ε, βάση του άρθρου 51 του κανονισμού περί κοινών συνεδριάσεων των Επιτροπών, που όπως γνωρίζετε παίρνει άδεια από τη διάσκεψη των Προέδρων και στις 26 Ιουνίου 2013 εδώ αυτή άδεια. Οι δύο λοιπόν εισηγητές των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας θα πρέπει να προτείνουν κοινή συνενέση, ένα ενιαίο σχέδιο έκθεσης, μία έκθεση δηλαδή, η οποία θα συζητηθεί σε κοινέ συνεδριάσεις, θα συζητείτε πάντα των δύο επιτροπών και κάθε κοινή συνεδρίαση θα έχει ειδική ημερήσια διάταξη. Το πλαίσιο της ενέργειας, της βιομηχανίας, του κλίματος, της ανταγωνιστικότητας είναι κάτι ε, το οποίο μας απασχολεί και ε, τις δύο επιτροπές και θέλουμε να αποφανθούμε για αυτά τα δύο θέματα. και θέλουμε να ανταλλάσσουμε απόψει σε αυτέ τι κοινέ συνεδριάσει για να μπορούμε να συνεννοούμαστε καλύτερα. Να βλέπουμε ο καθένα ε, το θέμα από τη σκοπιά του άλλου και να διευκολύνεται έτσι η δουλειά μα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και έχετε και πάλι το λόγο. Ωραία. Λοιπόν, ένα αρκτήριο λάκτισμα για την έκθεση και για τη συζήτηση. Έχουμε δύο συνεισηγητές ο Κόνατ Σιμάνσκι και η Άννη Τελβό από την Επιτροπή μας εναλλάξ για 10 λεπτά έχουν το λόγο οι συγητές, συνεισηγητές. Πρώτα από την Επιτροπή Βιομηχανίας ο κύριος Κόνατ Σιμάνσκι. Παρακαλώ. Ε, e, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για αυτή την ευγενική χειρονομία. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος αλλά καλεσμένο σας, παρακολουθώ τις εργασίες σας, οι οποίες επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα. Μαζί με την κυρία Ντελβό αποφασίσαμε να μην χωρίσουμε το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τμήματα κάποια για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, κάποια για την Επιτροπή Ενέργειας. Θα ασχοληθούμε με το έγγραφο συνολικά και οι δύο. Η ενεργειακή και κλιματική μας πολιτική μετά το 2020. Πώς θα είναι αυτή. Νομίζω πως καταρχάς πρέπει να δούμε τι καινούργια δεδομένα δημιουργεί αυτή η πολιτική, η οποία Δημιουργήθηκε πριν από λίγο καιρό η πολιτική στόχη, στόχη της πολιτικής ε, αυτής. Ήταν η εξή. Καταρχάς, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να διασφαλίσουν ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια και να συντελεστεί η κλιματική η ενεργειακή αλλαγή. Αποφασίστηκε λοιπόν να εισαχθεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και να εμπλουτιστεί η ενεργειακή χρήση με το 20% της ενέργειας να προέρχεται από τα ανανεώσιμες πηγές. Πιστεύω πως κανείς ε, δεν ε, διαφωνεί με αυτόν τον στόχο εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι κοινό πολιτικός ε, στόχος. Ο στόχος όμως αυτός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από το να θεωρούμαστε ενεργειακά αυτόνομοι. Πάνω από το 90% της ενέργειάς μας προέρχεται από ρηκτά καύσιμα και από το 2014 και μετά θα έχουμε οικονομικά προβλήματα στον τομέα αυτό. Προτάθηκε να γίνει μια έκθεση για την παγκόσμια κατάσταση. Σύμφωνα με την έκθεση, η γερμανική εθνική οικονομία δεν θα ανήκει πλέον στις μεγαλύτερες και πιο δυνατές οικονομίες του κόσμου και αυτή τη στιγμή γινόμαστε ολαιόνα και λιγότερο ανταγωνιστικοί. Ενεργειακή επάρκεια. Τώρα. Σε σχέση με το 1995... Έχουμε μειώσει βέβαια τις ε, εκπομπές ρήπων, όχι όμως ε, χάρη στην ενεργειακή μας πολιτική πιστεύω πως γι' αυτό ευθύνεται και η μείωση της ε, παραγωγής. Η παραγωγή χάλιβα, όπως είπαμε και χθε, είναι 30% κάτω από τις ε, δυνατότητες παραγωγής. Και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο λειτουργεί αυτό το σύστημα είναι η αγορά εκπομπών, η αγορά πιστοποιητικών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πολιτική πίεση στην αγορά αυτή και οι τιμές των πιστοποιητικών ανεβαίνουν τεχνητά. Έχει μειωθεί η ζήτηση και διορθώνονται ως αποτέλεσμα και οι τιμές των ε, πιστοποιητικών. Είναι αρκετά περίπλοκο το σύστημα, όμως πιστεύω αρκετά εξισορροπημένο. Δυστυχώς δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, κάνει διαφορετική προετοιμασία για την ε, ανάληψη του κόστους ε, των πιστοποιητικών. Το κόστος δεν είναι το ίδιο από χώρα σε χώρα, οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ίδιες, όπως επίσης και οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τώρα. Πολλές φορές εδώ υπάρχουν προβλήματα με την χρηματοδότηση, η οποία θα μπορούσε να είχε δοθεί σε, για παράδειγμα, στην έρευνα. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, οι φτωχότερες χώρες έχουν να αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, τα πιστοποιητικά για το φυσικό αέριο, τα κριτήρια αξιολόγηση για το φυσικό αέριο. Ε, επίσης υπάρχουν και οι βιομηχανίες που είναι πολύ απαιτητικές ενεργειακά, όπως για παράδειγμα η βιομηχανία του Χάλιβα. Ο κλάδος αυτός, όπως ε, είπα, έχει 30% λιγότερα πιστοποιητικά και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την παραγωγή χάλιβα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποσταθεροποιείται ο κλάδος στην Ευρώπη. Και αυτό έχει άμεσες συνέπειες και στην βαριά βιομηχανία λόγω του ε, βιομηχανικού κύκλου παραγωγής που πολλές αρχη διαρχεί 20-30 χρόνια. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ αρνητικό. Δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα για τη βιομηχανία και οι συνέπειες αυτής της πολιτικής απόφασης θα είναι επίσης αρνητικές. Γι' αυτό στην γνωμοδότησή μου συμπεριέλαβα ορισμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη Σίγουρα συμφωνούμε όλοι να μειώσουμε τις ε, εκπομπές ε, ρήπων. Η αλλαγή όμως αυτή πρέπει να γίνει σύμφωνα με την παγκόσμια κατάσταση. Να έχουμε και την παγκόσμια σύμφωνη ε, γνώμη. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εκτός από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βραζιλία και οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ινδία και η Κίνα είναι πάρα πολύ δυνατές βιομηχανίες και ο στόχος της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα πρέπει να είναι κοινό. Πρέπει λοιπόν να γίνει ανάλυση, να δούμε τι χρειάζεται εάν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές μέχρι το 2050. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερες αναλύσεις, λεπτομερέστερες αναλύσεις, ε, συγκεκριμένα για την κάθε χώρα και ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης η ανάπτυξη του ελεύθερου εμπορίου και το τονίζω αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης και την αιρεσιμότητα. Ας δούμε για παράδειγμα τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρέπει να δούμε τη συσχέτιση της ε, αμερικανικής βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σιμάνσκι. Κύριε Αντελβό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το άρθρο 51 και τον κύριο Σιμάνσκι που μόλις έκανε την δική του παρουσίαση για το κείμενο στο οποίο και ήδη δύο έχουμε αναλάβει οι ε, δεν θα ταυτίσω απολύτως τις απόψεις μαζί του. Πιστεύω ότι βρίσκεται ένα στα προδρόμια Ευρώπη σε σχέση με τι κλιματικέ τη δεσμεύσει, προκειμένου να δημιουργήσει μια νέα αγορά για την ενέργεια και για να μειώσει την ενεργειακή τη εξάρτηση, να ανακάμψει η οικονομία τη με πράσινε θέσει εργασία, να ξαναρχίσει η ανάπτυξη και να προωθήσει τι τεχνολογικέ λύσει με διάφορες καινοτόμους προτάσεις. Είναι πολλαπλές λοιπόν οι προκλήσεις και είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να δώσουμε αποκρίσεις διατομιακές ε, και ολοκληρωμένε, με διορατικότητα. Α είμαστε ρεαλιστέ. Ένα μόνο στόχο μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να υπάρξει, ε, συνδεδεμένο με την ε, τιμή του άνθρακα και την ουδέτερη τεχνολογία. Αλλά μπορεί μόνο αυτό να καλύψει το σύνολο όλων των προκλήσεων που προανέφερα. Επιτρέψτε μου να έχω τι αμφιβολίε μου. Διότι εδώ, το επαναλαμβάνω, έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με την απεξάρτηση από τον άνθρακα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστο, αλλά να δίνουμε ε, την ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία των ενεργειακών πόρων, να τονώσουμε την απασχόληση και τι θέσει εργασία, να μείνουμε σε ηγετικό ρόλο στην ε, τεχνολογία και στην ανάπτυξη. Αυτό και μόνο ο στόχο κατά την άποψή μου, θα ήταν συνώνυμος με ε, με παλινδρόμηση. Είναι κρίμα για τι τεχνολογίε που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα πρέπει όμω να συνεχίσουμε ακριβώ ε, στην ίδια οδό που το πακέτο για το κλίμα 2020 έχει προδιαγράψει. Όχι, πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματά μα σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του, τι ανεπαρκέ του, τι απλεψίε του, από κάποιε ασυνέπειε που υπήρξαν στο σχεδιασμό. Ήδη είδαμε από τα μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί σήμερα ότι υπάρχουν αρκετέ αδυναμίε, αλλά χρειάζεται επανεξέταση των όσων υπάρχουν. Και αυτό α γίνει χωρί δογματισμού, χωρί ιδεολογικέ προκαταλήψει, χωρί ε, να ξεχνάμε το ρεαλισμό και τον πραγματισμό που απαιτείται εδώ. Δηλαδή, ανοίγει συζήτηση, αυτό θέλω να πω, σε σχέση με τα σημεία κλειδιά που θα συμπεριλαμβάνει αυτή η έκθεση. Εγώ συνηγορώ υπέρ τη συνέπεια και τη συνέχεια να συνεχίσουμε μια προσέγγιση συνδυάζοντα τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Νομίζω ότι είναι τρία σημεία αξιοπιστία που απαιτούνται. Η προσέγγιση αυτή έχει τριπλό στόχο. Να υπάρξει καλύτερο συντενεσμό ε, όλων αυτών των στόχων με σκοπό να περιοριστεί το κόστο, αλλά ο καθένα από του στόχου να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένε προκλήσει, στοχευμένα και να αλληλοσυνδέονται προκειμένου να αλληλοενισχύονται. Θα πρέπει να διαλέξουμε μία επιλογή που να μην μας δημιουργεί ε, ε, ένα αρνητικό προηγούμενο για το μέλλον. No regrets option. Αυτές ε, οι λύσεις πολλές φορές βέβαια προκαλούν τις περισσότερες συζητήσει, είναι πιο αμφιλεγόμενες. Γιατί λοιπόν να επιλέξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις ε, συμβατικές πηγές ενέργειας, για να μειωθεί το κόστος της ενέργειας στο μέλλον, για να υπάρξει ένα καλύτερο μείγμα ενεργειακών πόρων στο μέλλον, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που να ε, μην είναι μόνο παροδικέ. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ο στόχος μας. Νομίζω το πρόβλημα είναι τα μέσα που θα επιλέξουμε, η οδό που θα επιλέξουμε για να καταλήξουμε εκεί. Γι' αυτό μέχρι τώρα ε, είναι όμοιρο η ενεργειακή αγορά όλων των προηγούμενων επιλογών μας. Χρειάζεται να στηρίξουμε και να επιδοτήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αυτό ήδη γίνεται σε κάποια κράτη-μέλη με καλύτερο συντονισμό και συνέπεια από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αυτό δεν υπάρξει υπάρχει πρόβλημα. Και είμαι πεπισμένη ότι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια μπορούν να είναι κερδοφόρε και μακροπρόθεσμα και δεν θα χρειάζονται πλέον επιδότηση. Εδώ πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ πράσινη ανταγωνιστική ενέργεια και πράσινη ενέργεια που ακόμα βρίσκεται σε στάδιο ορίμανση, οικειοπορία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ενεργειακή ενέργεια, θα πρέπει να αφήσουμε τι επιχειρήσει να λειτουργούν και να εξυπηρετούν του τελικού καταναλωτέ. Αυτό είναι περισσότερο από χρήσιμο προφανώ, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε και την ε, δική μα ε, αυτάρκεια την ενεργειακή. Ακόμα και με τη νέα οδηγία του 2014, αυτή που πρόκειται να ισχύσει το 2014, θα πρέπει να διατηρήσουμε τον πρωταρχικό μα σκοπό. Να μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να προσανατολιστούμε στα κριτήρια τη ε, κερδοφορία. Ε, Εξάλλου υπάρχει και κάποιο ενεργειακό πλεόνασμα κάποιες φορές που δεν έχει ε, καταναλωθεί. Όσο για τους δεσμευτικούς στόχους να πω ότι στη δέσμη μέτρων όπως παρουσιάζεται, οι μόνοι στόχοι που θα πετύχουμε είναι αυτοί που ήδη είχαν ε, θεωρηθεί δεσμευτικοί από την αρχή. Κάποιοι θα μου πούν ότι η πίεση μπορεί να δίνει αποτελέσματα. Όμω έχουν ε, μπλοκαριστεί και κάποιε επενδύσει, έχουν μειωθεί επενδύσει σε χαμηλή κατανάλωση άνθρακα προϊόντα. Όχι. Εδώ θέλουμε μία μη δεσμευτική προσέγγιση που να οδηγεί σε έναν ενιαίο στόχο. Ε, δεν γίνεται αυτό. Οι στοχευμένοι στόχοι, οι στοχευμένε προτεραιότητε μάλλον, δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε βιομηχανικό τομέα να προβλέψει τα κέρδη του και να ξέρει τι κάνει βιομηχανία όμω δεν κάνει τι πολιτικέ επιλογέ. Πρέπει να γίνει ένα τέτοιο σχεδιασμό των επενδύσεων, ώστε ο ιδιωτικό τομέα να μπορέσει μακροπρόθεσμα, με διορατικότητα, να αναπτύξει τα επιχειρηματικά του πλάνα. Πολλέ εταιρείε, πολλέ επιχειρήσει έχουν εκφράσει αυτή την επιθυμία. Προκειμένου να ξεπεράσει η Ευρώπη το σημερινό αδιέξοδο, θα πρέπει να έχει ένα σαφέ, ξεκάθαρο πρόγραμμα, εξεπιδετώντα την ανάπτυξη και επιτρέποντα τι επιχειρήσει να λειτουργήσουν σε ένα ασφαλέ πλαίσιο. Δεν θέλουμε αντιπαραγωγικέ λύσει. Το να έχουμε λοιπόν ένα όριο ε, δεσμευτικό ελληνικό μακροπρόθεσμα, σημαίνει ότι θα έχουμε και στόχους μετρήσιμους και ότι θα μπορούσαμε να αναλάβουμε και διευθυντικά μέτρα εφόσον χρειαστεί. Για τους ε, στόχους του 2015, λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ενδιάμεσοι στόχοι. Αυτό επιτρέπει μια γραμμική ανάπτυξη και μια ανακατανομή των ε, προσπαθειών μα στον χρόνο, προκειμένου να περιορίσουμε τον... την ένταση των επενδύσεων εφόσον χρειαστεί και να ανακατανεμηθούν ε, οι οικονομίες που μπορεί να γίνουν. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να έχουμε διατομιακέ διατάξει, να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα, να κοιτάξουμε την τιμή τη ενέργεια και την ασφάλεια τη προμήθεια και την ενεργειακή μα αυτάρκεια. Αυτά τα στοιχεία είναι καθοριστική σημασία και από την πλευρά των επιχειρήσεων και εταιριών αλλά και των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα προφανώς θα πρέπει να είναι ε, ένα νήμα που θα οδηγήσει την πορεία της έκθεσης. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Έχουμε και ένα δυναμικό ανάπτυξη στα χέρια μας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τέτοιες τεχνολογικές και οικονομικές λύσεις που το δυναμικό αυτό να το επιτρέψουν να προχωρήσει, να αξιοποιηθεί. Οι ειδικοί μας μιλάνε για την αύξηση της τιμής της ενέργειας που έχουν σχέση και με την αύξηση των αναγκών σε ενέργεια και με το μείγμα ενεργειών πόρων που, ενεργειακών πόρων που χρησιμοποιούμε. Αυτό θα βελτιωθεί πολύ ω οποίο εφόσον χρησιμοποιήσουμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Επιμένω πολύ σε αυτό. Χρειάζονται λύσει, ε, backup για τα κράτη-μέλη και συγκεκριμένε ειδικέ ενεργειακέ συνταγέ ανάλογα με τι ανάγκε του καθένα. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τι τιμέ τη ενέργεια προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκε τη Ένωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ω προ την ασφάλεια τη προμήθεια, την προστασία και την αυτάρκεια, το να μειωθεί η εξάρτησή μα και να διαφοροποιηθούν οι πηγές τροφοδότησής μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε τους αριθμούς των Ένωση, η Ένωση είχε τουλάχιστον 250 δις εισαγωγές ορεικτών καυσίμων την περσίνη χρονιά. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν όρια μακροπρόθεσμα για μια ενιαία ενεργειακή αγορά προ την οποία πρέπει να οδεύσουμε στο δυνατόν ταχύτερα. Με διασυνδέσει, με δίκτυα, με την πρόοδο τη πράσινη τεχνολογία. Μπορούμε να μειώσουμε το έλλειμμα του εμπορικού μα ισοζυγίου, του ενεργειακού εμπορικού μα ισοζυγίου, κάτι που είναι σημαντικό γιατί το 2012 το εμπορικό μα ισοζύγιο έδειχνε 483 δις ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν στην έκθεση αυτή να ε, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο δυναμικό των καταμελών, στην κατανομή των προσπαθειών μεταξύ των καταμελών και την ε, ε, μεγαλύτερη προσοχή στις βιώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Θέλω να έχουμε έναν πλούσιο διάλογο για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και όλες τις τυχές και ελπίζω ότι θα είναι παραγωγικός αυτός ο διάλογος και όλη η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντελβό. Πάμε. Σκιώδης ηγητές τώρα. Ε, πρώτα από την Επιτροπή ε, βιομηχανίας, μετά περιβάλλοντος, εναλλάξ, να είστε σύντομοι για να μπορέσουμε όμως να ανταλλάξουμε απόψεις όλοι, να πάρουν όλοι το λόγο. Χέρμπερτ Ρόιλ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν θέλει. Μα εδώ σε λέει ότι είσαι σκιώδης. Δεν θέλει. Καλά. Η κυρία Ουλφσκοκ από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Όδηση ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, ξέρουμε ότι το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές, το πρόγραμμα σύντομα θα δημοσιευτεί. Υπάρχουν πολλές νέες δυνατότητες που ανοίγονται χάρη σε αυτή την έκθεση και βάσει των όσων λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πάνελ που θα δημιουργηθούν για τις συζητήσεις περί κλίματος, ήδη θεωρούν ότι το 90% του πλανήτη θα υποστεί τις συνέπειες της υπερθέρμανσης. Η υπερθέρμανση αυτή κυρίως οφείλεται στην ανθρώπινη δράση και δραστηριότητα. Εν μέρη στην αύξηση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα που έχουν οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και μάλιστα σημειώνεται ότι εδώ και 800 χρόνια δεν υπήρχε τόσο διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Θα διατεθούν λοιπόν όλα αυτά στην κοινή γνώμη και σίγουρα αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι όλο και λιγότερο λιγοστεύει ο χρόνος που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές με διαφορετικές καταστροφικές συνέπειες ανά περιοχή του κόσμου. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η χρονική συγκυρία. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που έχουμε σε επίπεδο ομάδων. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η ευθύνη που έχουμε αναλάβει είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι από κοινού να βρούμε μια λύση που να είναι αποδεκτή όχι μόνο για μας αλλά για όλον τον πληθυσμό του πλανήτη και επίσης για τις μελλοντικέ γενιές. Όπως είπατε, χρειάζονται εδώ ε, Περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρειάζεται περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, οι τιμές είναι ήδη πολύ υψηλές προσωπικά. Εγώ και τα περισσότερα μέλη της ομάδας μου δεν βλέπουμε να υπάρχει άλλη επιλογή. Θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει πλειοψηφία που να στηρίξει τους δεσμευτικούς στόχους. Εάν έχουμε δεσμευτικούς στόχους, τότε μπορεί τα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη της Ένωσης να μπορέσουν να εξεύρουν την πλέον ταχεία και την ευστοχότερη λύση για να πετύχουμε από κοινού αυτούς τους στόχους. Εάν δεν έχουμε δεσμευτικούς στόχους, δεν θα προστατεύσουμε παρκώς τους πόρους μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στην ομάδα μου, όπως έχουμε συζητήσει μάλλον στην ομάδα μου, και πιστεύω να συμφωνήσουν και άλλοι συνάδελφοι ότι πρέπει να υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο ορισμό για όλα αυτά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε φτηνέ λύσει. Θα πρέπει να επιδιώξουμε την τόνωση των επενδύσεων. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την αποθήκευση, με την διανομή, την παραγωγή της ενέργειας. Όλα αυτά είναι προφανώς ε, καθοριστική σημασίας για μια αγορά ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Για συγκεκριμένους τομείς, όπως το πετρέλαιο, προφανώς σημαντικό είναι να ορίσουμε στόχους ε, ως προς το ως προς το σημείο αυτό, αν θέλουμε να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα, θα πρέπει να έχουμε υψηλότερες φιλοδοξίες. Θα πρέπει να λάβουμε σαφείς αποφάσεις και να ορίσουμε συγκεκριμένους στόχους. Επιπλέον, θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε και το σύστημα φορολόγησης της ενέργειας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην δεχόμαστε σε αυτό το επίπεδο την ε, ανάλυση που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρξει φορολογία για την ενέργεια που να λαμβάνει υπόψη και την ενέργεια, τη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται και την περιεκτικότητα σε διοξίδιο του άνθρακα. Θα πρέπει αυτά να οριστούν με τρόπο όσο το δυνατόν σωστότερο εξ αρχής και όχι διαρκώς να διορθώνουμε τα πράγματα εκ των υστέρων αφού προκύψει μια καταστροφή. Υπάρχουν και άλλες πηγές ενέργειας. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο ενδοτικοί στην ε, προσέγγισή μας. Θα πρέπει να βρούμε το καταλληλότερο σύστημα, να δούμε τι γίνεται σε περιπτώσεις διαρροών λόγου χάρη. Θα πρέπει να δώσουμε βάρος σε αυτά που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό, γρήγορα και να μην ξεχνάμε τι γίνεται και με τα βιοκαύσιμα. Ε, αναμένω και εγώ τι απόψει των συναδέλφων. Ευχαριστώ, Τόμσον. Από σοσιαλιστέ και δημοκράτε και όδηση γήτρια στην ε, Επιτροπή Βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε 355 δισεκατομμύρια ευρώ για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων. Επαναλαμβάνω, 355 δισεκατομμύρια. Είναι περίπου το ετήσιο ΕΠ της Πολωνίας. Πολωνία ολόκληρη. Μια Πολωνία το χρόνο πληρώνουμε για να ε, φέρνουμε ορυκτά καύσιμα στην Ευρώπη. Περίπου το 60% του φυσικού αερίου και 85% του πετρελαίου και περίπου το μισό άνθρακα εισάγουμε. Σύμφωνα με την Διεθνή ε, Υπηρεσία Ενέργειας θα αυξηθούν αυτά το 2035. Αυτά τα στοιχεία τα αριθμητικά έχουν σημασία όχι μόνο στη μεγάλη συζήτηση που κάνουμε για την ενεργειακή εξάρτηση, αλλά και για την τιμολόγηση της ενέργειας. Ορισμένοι αρέσκονται στο να συγκρίνουν τις τιμές στη Ρωσία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και να το χρησιμοποιούν ε, ως επιχείρημα για λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές ε, για το κλίμα και την ενέργεια στην Ευρώπη. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το κλίμα και η ενέργεια παίζουν μικρό ρόλο στη τιμολόγηση της ενέργειας. Οι γεωλογικές ε, καταστάσεις στις Ηνωμένε Πολιτείες και στη Ρωσία και ε, τα μορφώματα γενικότερα είναι διαφορετικά από ό,τι στην Ευρώπη. Εμείς εισάγουμε ορεικτά καύσιμα, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ρωσία είτε έχουν φυσικούς πόρους, ε, ή γίνονται ανεξάρτητοι γιατί παράγουν ενέργεια. Επίσης, η σημερινή τιμή εμπορίας εκπομπών ETS είναι τόσο χαμηλή που είναι λιγότερο από 5% του μέσου τιμολογίου της ενέργειας στην Ευρώπη και επίσης ε, πολύ μικρό κλάσμα του συνολικού κόστους είναι ε, βασικά η εξάρτηση από τις αγωγές κυριαρχεί και όχι η πολιτική για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρόσφατα έκανε μια μελέτη που λέει ότι η κλιματική νομοθεσία δεν σήμαινε επιπλέον κόστος το 2012 για τις περισσότερες χαλιβουργίες στην Ευρώπη. Παρόλο που συμφωνώ ότι οι τιμές ε, μπορεί να είναι πρόβλημα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, εμείς νομίζω εστιάζουμε στους λάθος παράγοντες όταν προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Κανονικά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τα τεράστια ποσά που δαπανούμε για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων πρακτική λύση. Δεν είναι και τόσο δύσκολη. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους και οράματα για το μέλλον, για την εξέλιξη και τον εξυγχρονισμό του ενεργειακού μας τομέα. Το 2030 θα πρέπει να έχουμε δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακή απόδοση, οικονομία δηλαδή, για να έχουν την ασφάλεια και οι επενδυτές και η βιομηχανία. Το 2007 Επτά, ε, ήδη είπαμε ότι θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους επενδυτές, στη βιομηχανία. Άρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι δεσμευτικούς στόχους. Και κατάφερε κανείς ε, από το 2007 τότε να πείσει μέχρι και το ε, Ζακ Σιράκ και τους ίδιους τους Πολωνούς για αυτό το θέμα. Ε, μια ευρωπαϊκή στατηγική χρειάζεται για να μειωθεί η εξάρτησή μας από τις εξαγωγές. Γιατί ποιος κερδίζει, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ο Πούτιν και η Γκάσπρομ τελικά από όλη αυτή την ενεργειακή μας πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Φιώνα Ευχαριστώ πολύ. Σημείωσα αυτά που είπε η κυρία Ούλφσκοκ για την ε, έκθεση περί κλιματικής αλλαγής και όντως αυτό είναι το πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Ας θυμόμαστε όμως ότι το πακέτο αφορά τόσο το κλίμα όσο και την ενέργεια και η κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο αιώνας μας. Αλλά ας αφήσουμε λίγο την κλιματική αλλαγή και ας δούμε τις ενεργειακές επιτυχίες αυτής της έκθεσης, διότι είναι σαφές από όλα όσα συζητήσαμε σήμερα και προηγουμένως στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ότι, ότι και τα κράτη-μέλη και η πολιτική σήμερα ασχολούνται με τα θέματα της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας. Ας αρχίσουμε λοιπόν από αυτά και ας δούμε τι κάνουμε και τι θα κάνουμε από εκεί και στο εξής. Όσον αφορά το τι θα κάνουμε από οικονομικής ε, πλευράς, η απάντηση είναι προφανής, πιστεύω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε περισσότερο ενεργειακά αυτάρκεις. Αυτό μας κάνει και οικονομικά αυτάρκεις. Και είναι ενδιαφέρον το ότι υπάρχει τώρα μία έκθεση για ενεργειακή αυτάρκεια στα πλαίσια της οικονομικής ε, αυτάρκειας. Διαφορετικά, αν σπαταλούμε ενέργεια, είμαστε και οικονομικά αφαιρέγγι. Υπάρχουν, όπως είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, αν χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια, βοηθάμε και την τοπική οικονομία. Εξοικονομούνται χρήματα, ιδιαίτερα σημαντικό αυτό σε καιρούς κρίσης και αντιμετωπίζεται η φτώχεια. Εκτός από αυτό, οι μικρές επιχειρήσεις γίνονται και πιο ανταγωνιστικές, διότι δεν χρειάζεται να πληρώσουν ένα τεράστιο ποσό για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Από πλευρά ε, λοιπόν ε, αυτάρκειας και ανταγωνιστικότητας πρέπει να αρχίσουμε πρώτα να, δούμε, να βλέπουμε τι γίνεται με την ενεργειακή αυτάρκεια και να μην κοιτάζουμε τα επιμέρους τμήματα της ε, νομοθεσίας, να μην αποσπο... αποσπάται η προσοχή μας από αυτά. Τώρα, τι γίνεται για με το μείγμα της ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μεγάλο άγχος σχετικά με την ενέργεια και ανεξαρτησία. Και φυσικά η... ο πλούτος ε, ενέργειας που έχουμε είναι ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και αυτό μας κάνει και ανταγωνιστικούς. Ο τομέας που έχει σημειώσει ανάπτυξη σε περίοδο κρίσης και ο τομέας στον οποίο ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώ ε, κινδυνεύει να χάσει αυτή την ηγετική θέση, είναι οι ανανεώσιμε. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, πηγέ που έχουμε στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το σχιστολιθικό αέριο, το οποίο ίσως είναι μόδα Ίσως σε μερικά χρόνια αναρωτιόμαστε γιατί τόσο ντόρος με αυτό το πράγμα, όπως και με τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Το πρόβλημα όμως της κλιματικής αλλαγής παραμένει και εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της ε, κλιματικής αλλαγής. Ας αναλογιστούμε λοιπόν εάν η βιομηχανία μας χρειάζεται το σύστημα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Τώρα, όταν κοιτάζουμε τους εγγυγενείς επόρους, όπως είπα, βλέπουμε πάντα πως έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό είναι κάτι ανεξάντλητο. Δεν μπορεί κανείς να μας πάρει τον αέρα που έχουμε. Στην Βόρεια Θάλασσα έχουμε τις μεγαλύτερες ε, εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας στον κόσμο και πιστεύω πως όσο περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχουμε, τόσο περισσότερο ενεργειακά αυτάρκης θα, θα είμαστε. Αυτά από πλευράς ανταγωνιστικότητας και ενεργειακής αυτάρκειας. Εμείς, συμπεραίνω, είναι πάρα πολύ λογικό να επικεντρωθούμε σε αυτά. Τώρα, όσον αφορά τι επιχορηγήσει ε, για τι ανανεώσιμε ε, πηγέ ενέργεια, ορισμένοι είπατε πω ε, μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από το τι πήγε στραβά με αυτό. Βέβαια, κύριε Σιμάνσκι, επειδή το αναφέρετε εσεί, να πω ότι ορισμένε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι πάρα πολύ καινούργιε. και ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο τη έρευνα και πρέπει να τι αναλύσουμε περισσότερο. Πρέπει να προχωρήσει η τεχνολογία και δεν πρέπει λοιπόν να τους εμποδίσουμε, να εμποδίσουμε την έρευνα, εμποδίζοντας και την ε, χρηματοδότηση. Και τώρα όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου, η στάση μας δεν διαφέρει και πολύ από την στάση της Κομισιόν. Υπάρχει έμφαση στις ε, ανανεώσιμες πηγές. Υπάρχει αυτή η τακτική του no regrets. Και πιστεύω πως ε, κοιτάζουμε το πράγμα από λάθο σκοπιά. Αν δούμε πρώτα τι γίνεται με την ενεργειακή αυτάρκεια και μετά ασχοληθούμε με το σύστημα εμπορίας εκπομπών, θα βοηθήσουμε τη βαριά βιομηχανία μας, διότι η βαριά βιομηχανία μας θα χρειάζεται λιγότερα πιστοποιητικά ETS, ε εάν βασιστεί περισσότερο σε ανανεώσιμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Γκερμπράντι μίλησε από το στόμα. Εκπροσωπήθηκε από εσά. Η κυρία Σάτου χάσει και μετά ο Πάσα Χάουτ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απολύτως με τη Μαρίτα Ούτσκοκ, την κυρία Τόψεν και την κυρία Χολ για την ανάγκη να μην έχουμε ένα μόνο στόχο ε, ε, του θερμοκηπίου, αλλά τρεις στόχους, τις ανανεώσιμες και την ενεργειακή απόδοση. Ε, να πω όμως κάτι για την κλιματική αλλαγή την ίδια. Γνωρίζουμε ότι αύριο η IPCC θα εκδώσει την επόμενη έκθεσή τους. Τι έχει δημοσιευθεί ήδη όμως και από τη UNED και την Παγκόσμια Τράπεζα γνωρίζουμε το εξής. Εάν δεν επιταχύνουν τις προσπάθειές του υπέρ του κλίματος οι χώρες στον κόσμο, είναι πιθανό να αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη ακόμα σε αυτό το αιώνα κατά 3 με 4 βαθμούς. Και τελικά μπορεί να έχουμε ένα κλιματικό σύστημα το οποίο είναι πολύ πιο πέρα από αυτό που έχει ζήσει η ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια του ανθρώπινου πολιτισμού στη γη, 10.000 χρόνια δηλαδή. Αν συνεχίσουμε με την παρούσα τακτική σημαίνει ότι στέλνουμε τα παιδιά του σήμερα και τα βρέφη σε έναν άγνωστο πλανήτη, σε ένα πλανήτη που δεν θα ξέρουμε πώς θα ζούμε, δεν μπορούμε να το δεχόμαστε αυτό. Φανταστείτε να έρθει ένας εξωγήινος να παγάγει τα παιδιά μας και τα βρέφη μας, να τα πάει σε άλλο πλανήτη. Πώς θα αντιδρούσαμε. Δεν θα ρωτούσαμε πόσο κοστίζει ε, κιλοβατόρα, ένα λεπτό ή δέκα λεπτά παραπάνω. Πόλεμο θα του κάναμε αυτόν που θέλει να παγάγει τα παιδιά μας. Και αυτό ε, αφορά την κλιματική πολιτική και δεν το καταλαβαίνουμε. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ήδη ε, την τιμή ε, που πληρώνουμε το τίμημα για την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πάντα θα πρέπει να είναι τμήμα της συζήτησης για το κόστος, για την κλιματική πολιτική. Και όπως ε, ήδη ανέφεραν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας υπολογίζει ότι θα αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου στο μέλλον και πολύ περισσότερο ε, από ό,τι υπολογίζει η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή στη Βίβλο για το 2030. Για τη χώρα μου, τη Φινλανδία, όπου η βιομηχανία χάρτου ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα ο βασικός κλάδος της οικονομίας, εισάγουμε ρηκτά καύσιμα, πληρώνοντας το ίδιο τίμημα με αυτό που εισπράττουμε για την εξαγωγή χάρτου. Δηλαδή είναι για μας μεγάλη δαπάνη. Και ε, γενικότερα ε, ο τομέας αυξάνεται από το 2008 μέχρι το 2011. Δηλαδή μετά τη ε, οικονομική κρίση, η καθαρή τεχνολογία έχει διπλασιαστεί, το clean tech. Μετά το διαδίκτυο και το τζόγο ή το τζόγο στο διαδίκτυο μάλλον είναι η βιομηχανία που αναπτύσσεται με τους ε, ταχύτερους ρυθμούς. Πέρσι είχε ένα ποσοστό ανάπτυξη 15%. Είναι ρεαλιστικό λοιπόν να σκεφτόμαστε ότι μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα ε, μπορεί να συνδυαστεί και θα συνδυαστεί με την ανταγωνιστικότητα στην οικονομία. Και ένα τελευταίο σημείο. Πολύ συχνά ακούτε ότι η Ευρώπη είναι μόνη της σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ισχύει απλούστατα αυτό φέτος. Η Κίνα άρχισε να κάνει εμπορία εκπομπών στο σημαντικότερο τμήμα της οικονομικάς, τη μεγαλύτερη και την πιο δραστήρια περιοχή της και είπε ότι θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα το σύστημα εμπορία εκπομπών. Μόλις πριν από λίγε μέρες η κυβέρνηση του Πρόεδρου Ομπάμα στην Αμερική αποφάσισε να ε, ε, εισαγάγει πρότυπα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρότυπα και πρωτογραφές που εμεί δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που αν κατάλαβα καλά σημαίνουν ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν νέα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια χωρίς ε, δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Θα είναι παράνομη η λειτουργία τους πλέον στην Αμερική. Και όταν μιλούμε για την παγκόσμια εικόνα θα πρέπει να καταλαβαίνουμε και να βλέπουμε και τα θετικά, όχι μόνο τα αρνητικά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενθαρρύνουμε και να δίνουμε το καλό παράδειγμα για τις θετικές εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Σιμάνσκι. Mm, Ήθελα και εγώ να πιστήσω την προσοχή σας στους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ μιλάμε για αξιοπιστία και είναι πολύ σημαντικός ο όρος αυτός. Αξιοπιστία. Διότι το θέμα είναι έναντι ποιου πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιόπιστη. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε αξιόπιστοι ενώπιον των ε, βασικών μας εταίρων που συμμετέχουν μαζί μας στον αγώνα για την αναχέτηση των ε, κλιματικών αλλαγών της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στην ε, διάσκεψη της Βαρσοβίας για το κλίμα θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ίσως και μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Έχουμε στόχους αμφιλεγόμενους και πολλές φορές αντιφατικούς. Ε, πρόσφατα ο πρόεδρος Ομπάμα στην, ε, στο διάγγελμα του προς το έθνος είπε ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και ο περιορισμός των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα έχει να κάνει με την επιβίωση του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ενεργειακή ασφάλεια και η διασύνδεση των δικτύων είναι ο σωστός δρόμος. Να μην ξεχνάμε εδώ και τη σημασία της οικονομίας καθώς συζητάμε με τους εμπορικούς μας εταίρους σήμερα. Έχει μετατοπιστεί η παραγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες με χώρες που οι στόχοι τους και οι φιλοδοξίες τους για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ χαμηλότερα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να έχουμε στόχους φιλόδοξους. Δεν είναι όμως το ζήτημα να έχουμε μόνο οικολογικούς στόχους και προτεραιότητες για να σώσουμε τον πλανήτη. Όχι. Χρειαζόμαστε περισσότερη σημασία, περισσότερες περισσότερη τόνωση της ευρωπαϊκής μας οικονομίας. Γι' αυτό μίλησα για την αξιοπιστία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντική η σταθερότητα και η συνέπεια. Γι' αυτό ε, θέλουμε να συνομιλήσουμε και με εκπροσώπους της βιομηχανίας. Και γι' αυτό το θέμα αυτό τους απασχολεί διακαώς και τους ίδιους. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τον περιορισμό των δικαιωμάτων ε, εκπομπών και την ανταλλαγή τους και γι' αυτό ασχολείται και με το τι κάψιμα χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και τι μεταφορικά μέσα επιλέγονται. Εδώ μιλάμε για πολύ σημαντικά κονδύλια. Κονδύλια τα οποία ε, τα επενδύει θέλει να έχει και τη βεβαιότητα ότι θα αποφέρουν κέρδη τα χρήματά του. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό για το βιομηχανικό και τον επιχειρηματικό κόσμο να θυμίσω ότι πρόσφατα στην ε, Επιτροπή μας ήρθε και ο Υπουργός ε, που μας μίλησε για την σημασία των διεθνών συμφωνιών και τις διαπραγματεύσεις και το πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Αυτό όμως δεν πρέπει να το βλέπουμε ε, ως ε, ένα τετελεσμένο γεγονός. Είναι η περίπτωση του ενός καλλιδονιού που δεν φέρνει την άνοιξη. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι είμαστε μεν ένα πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά οι δικές μας δράσεις μόνες τους δεν κάνουν τίποτα. Έχουμε να κάνουμε με μεγάλες οικονομίες, με γίγαντες απέναντί μας. Είχαμε ένα θα είχαμε μάλλον ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα ως προς την μείωση των εκπομπών, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο στο μέλλον, εάν ήταν διαφορετική στάση και οικονομική προσέγγιση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν η έκκληση που απευθύναμε στον κόσμο μπορούσε να εισακουστεί. Πρέπει να φτάσουμε σε συμφωνία. Ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ μας στις δικές μας συζητήσει, αλλά ακόμα πιο δύσκολο θα είναι να συμφωνήσουμε στο να έχουμε ευρωπαϊκή οικονομία με πολιτική βαρύτητα σε σύνοδο κορυφής για το κλίμα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε όλα αυτά να προχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χέρμπερτ Τρόιλ για το τέλος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλα όσα υπόθηκαν και θα προσπαθήσω τώρα να παρουσιάσω ορισμένα επιχειρήματα που θεωρώ σημαντικά. Είμαστε δύο επιτροπές και έχουμε το έργο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για ένα πάρα πολύ δύσκολο και περίπλοκο θέμα. Αυτό θα το καταφέρουμε μόνο εάν πραγματικά έχουμε μια εις βάθος ανταλλαγή απόψεων, εάν εργαστούμε στενά και πολύ. Ο κάθε ένας φυσικά έχει τη δική του προσέγγιση, ο κάθε ένας έχει τις δικές του προτιμήσεις. Όμως εάν επιμείνουμε σε προσωπικές απόψεις δεν θα προχωρήσουμε. Και μετά ας μην ξεχνάμε έχουμε και τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Στην αρχή έγινε λόγος για την ενεργειακή αυτάρκεια και την μείωση των εκπομπών και την κλιματική αλλαγή ως ε, η σημαντική στόχη μας. Και αυτό θα το καταφέρουμε μέσω του ενεργειακού μείγματο. Ένα άλλο συνάδελφο είπε ότι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων. Αλλά πραγματικά πιστεύετε ότι αυτές τις διαφορετικές απόψεις μπορούμε να τις υλοποιήσουμε μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που έχουμε έτσι ώστε να λάβει χώρα αυτή η ενεργειακή αλλαγή ούτε σε 100 χρόνια ή μπορεί σε 100 χρόνια, πάντως όχι μέχρι το 2030. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικές ε, διαφορετικές συνθήκες χρήσης της ενέργειας και οι στόχοι αυτοί θα έχουν διαφορετικές επιπτώσεις από κράτος σε κράτος και προτού, ε, θα έλεγα, προτού μιλήσετε για τρεις διαφορετικούς ε, στόχους Α δούμε καλύτερα τι μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και τι επιπτώσεις είχαν αυτά τα μέτρα. Έχουμε θέσει κάποιους στόχους για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και πιστεύω πως είμαστε σε καλό δρόμο. Θα τους επιτύχουμε, αλλά ας δούμε λίγο και τους ε, στόχους μας για τις ανανεώσιμες πηγέ ενέργειας. Εδώ τους στόχους αυτούς μπορούμε να τους ε, φτάσουμε, να τους ξεπεράσουμε κιόλας. Αλλά σας παρακαλώ να κοιτάξετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που θα προκύψουν εάν προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και τους τρεις στόχους αυτούς μαζί. Προσπαθήστε, προσπαθήστε να δείτε τι θα γίνει με το κόστος. Θα αυξηθεί το κόστος πάρα πολύ. Και οι κυβερνήσεις θα έχουν το δύσκολο έργο να εξηγήσουν στους ε, πολίτες τους γιατί θα πρέπει να ανεβάσουν τις τιμές. Όλοι φυσικά ε, εργαζόμαστε με στόχο την ε, ενεργειακή ενιαία αγορά, αλλά πραγματικά υπάρχει αυτή. Υπάρχει μια ενεργειακή ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε να υπάρχει. Τώρα, ενεργειακή αυτάρκεια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε τους στόχους. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε δεν μπορούμε. Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική άποψη και διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικούς στόχους. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση και από την άλλη κάνουμε λόγο για έξυπνα μέσα. σε κάποιε ε, χώρε ε, δεν υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι, υπάρχουν κίνητρα και αυτά έχουν αποδειχθεί πολύ πιο επιτυχημένα από οποιονδήποτε δεσμευτικό στόχο. Εσείς ε, εκπρόσωπος ε, του Ηνωμένου Βασιλείου κάνετε λόγο για ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά για θυμηθείτε τι έγινε πέρυσι που ψηφίσατε. Τι ψηφίσατε, πώς ψηφίσατε με το... και τι έγινε με το Συμβούλιο. Εντάξει, καταλαβαίνω εδώ από που προέρχεστε, όμως... Εάν θέλουμε να επιτύχουμε αυτού ε, τους στόχους χωρί τα ανεπιθύμητε παρενέργειες, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να δούμε εάν μπορούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους ακολουθώντας διαφορετική προσέγγιση, διαφορετική τακτική. Δεν είμαι... Δεν έχω καταλήξει σε κάποια απάντηση, δεν είμαι έτοιμος, όμως πιστεύω ότι αυτό που λέτε δεν είναι έξυπνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τα τρία πράγματα ταυτόχρονα. Δεν νομίζω πως είναι λύση, αμφιβάλλω γι' αυτό. Άκουσα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέροντα επιχειρήματα από συναδέλφου πολύ, ε, πολύ ενδιαφέροντα κριτήρια, ότι πρέπει να ε, είναι ρεαλιστικοί οι στόχοι, πρέπει να αυξήσουν την ε, ανταγωνιστικότητα, πρέπει να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες που έχει το κάθε κράτος μέλος και θα έλεγα ας σταθούμε σε αυτά, ας δούμε αυτό, αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και ας τα αναλύσουμε. Πραγματικά πιστεύω πως δεν είναι η καλύτερη λύση να, να, βάζουμε δύο καρπούζια κατά από την ίδια μας χαλιτρία στην προκειμένη περίπτωση. Ας ιεραρχήσουμε τους στόχους μας, ας δούμε τι θέλουμε πρώτα απ' όλα και τους επόμενους στόχους ας τους χρησιμοποιήσουμε ως τα μέσα για την επίτευξη του κύριου στόχου και έτσι και το Συμβούλιο στο τέλος θα συμφωνήσει μαζί μας. Διαφορετικά δεν έχει νόημα έτσι όπως το κάνετε αυτό τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόιλ. Με εσά φτάσαμε στο τέλος των παρουσιάσεων των σχεδόν εισηγητών. Όπως είπατε, πολλά θέματα της ενεργειακής πολιτικής στην αρμοδιότητα των κρατών ε, μελών. Είναι θέμα εθνικό. Αλλά δεν έχουν καταλάβει όμως επίσης πάρα πολύ ότι είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Τώρα, περνάμε στον δεύτερο γύρο. Ο Γιώ Λάινεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να πρόκειται για προστασία του κλίματος κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι το μοναδικό μας μέλημα. Υπάρχουν και μια σειρά άλλων σημαντικών θεμάτων, ασφάλεια στον ανεφοδιασμό. Ο κύριος Σιμάνσκι και άλλοι εξέφρασαν τη λύπη τους που εξαρτάται τόσο πολύ η Ευρώπη από εισαγωγές ενέργειας. Επίσης πρόκειται για νέους κλάδους της βιομηχανίας, είναι και βιομηχανική πολιτική, τεχνολογίες και που μπορεί να αναπτύξει κανείς. Επίσης και τελικά πρόκειται και για οικονομική ανάπτυξη. Ακριβώς ε, στην Ήπεθρο ή σε περιφέρειες απομακρυσμένες, νησιά, ε, όπου η ντόπια χώρια παραγωγή έχει ακόμα μεγάλο πεδίο να αναπτυχθεί. Και η πολιτική για το 2030 θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλο αυτό το πλαίσιο και όχι πολύ στενά την προστασία του κλίματος. Ο Κόρα Τσιμάνσκι είπε επίσης ότι το πρώτο πακέτο για το κλίμα από το 2008 είναι ακόμα πολύ νεαρό, αλλά έχει περάσει μια πενταετία. Μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να διαπιστώσουμε ότι είμαστε σε μια επιτυχημένη οδό θα επιτύχουμε το στόχο για το διεξίδιο του άνθρακα, 20% ανανεώσιμες και αφού έχουμε κάνει και ε, δεσμευτικό το στόχο για την ενεργειακή απόδοση, θα φτάσουμε και εκεί στο 20% εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή επιτυχίες έχουμε και ας μην τα περιγράφουμε όλα μαύρα. Και όσοι επένδυσαν εκεί ε, πραγματικά έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους ότι μπορούν να εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται. Έχουν ε, δημιουργηθεί πολλοί κλάδοι και στις ανανεώσιμες και στην εξοικονόμηση ενέργειας και αγαπητέ Χέρπερτ Ρόιλ, θα ήταν τώρα ανόητο τουλάχιστον να ε, στρίψουμε το τιμόνι προς την άλλη κατεύθυνση, στα μισά του δρόμου. Η κλιματική αλλαγή και η προστασία του κλίματος αντιμετωπίζεται, ναι, και χωρίς ενεργειακή απόδοση και χωρίς ανανεώσιμες, μπορεί να την κάνει κανείς και με πυρηνική ενέργεια. Και με άνθρακα, συνδέσμευση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Και υπάρχουν και σημαντικά συμφέροντα που το πάνε προς τα εκεί. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Είναι τεράστια η πίεση των λόμπι να δημιουργηθούν και να χτιστούν και άλλα πυρηνικά εργοστάσια. Και ο άνθρακας να δείτε τι λόμπι έχει. Δυστυχώ δεν γίνεται η δέσμευση και η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά προσοχή, προειδοποιώ. Αυτοί οι δύο υποστόχοι, οι δεύτεροι στόχοι, οι ανανεώσιμες και εξοικονόμηση ενέργειας, να μην ε, απεμποληθούν, διότι πηγαίνουμε ευθεία ε, στα μεγάλα εργοστάσια που είναι ο λεγόμενος καθαρός άνθρακας, αν συμφέρει με το CCS και τα πυρηνικά εργοστάσια. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε λίγο το σύστημα γιατί βλέπω ένα πρόβλημα στο ETS, το σύστημα εμπορίας εκπομπών, όσο περισσότερες ανανεώσιμες έχουμε και ενεργειακή απόδοση, τόσο λιγότερα είναι τα πιστοποιητικά. Κάτι τρέχει εκεί. Πώς θα το διορθώσουμε. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε με ε, τεχνητή άνοδο της τιμής ε, γιατί θα καταρρεύσει το σύστημα. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Θέλουμε μια Ευρώπη που να εξοικονομεί πόρους αλλά γι' αυτό χρειάζομαστε ένα τριπλό στόχο και όχι έναν απλό. Ευχαριστώ. Ξέχασα να πω ότι έχετε δύο λεπτά χρόνο αγόρευσης αλλά θα πρέπει να εξισορροπούμε και τις επιτροπές ε, Ήτρε, Ένβη και τις πολιτικές ομάδες. Η κυρία Γιόρδαν Σίσελη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ρόιλ. Όταν συζητούμε αυτό το θέμα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή. Αλλά Θέλουμε επίσης και να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το πρόβλημα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Ισχύουν αυτά που είπε ο Γιολάινεν. Αλλά η ανταγωνιστικότητα δεν λειτουργεί στον τομέα της ενέργειας. Στον τομέα της ενέργειας ε, σχεδόν καμία επένδυση δεν είναι ανεξάρτητη. Όλες είναι επιδοτούμενες. επιδοτούμε την αγορά φυσικού αερίου, την αγορά ορεικτών καυσιμών για να κρατήσουμε ανταγωνιστική την βιομηχανία. Ας έχουμε υπόψη τη λειτουργία της αγοράς, τις βασικές αρχές της λειτουργίας της αγοράς. Πιστεύω πως χρειαζόμαστε μεν το ETS, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν τόσες μεγάλες επιδοτήσεις. Το σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί. Πρέπει να έχουμε έναν ενιαίο στόχο και ο στόχος αυτός είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δεν λέω βέβαια να καταργήσουμε τελείως τις επιδοτήσεις, αλλά να επενδύσουμε και στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν έχουν αρκετές, αρκετή χρηματοδότηση ακόμα. Χρειαζόμαστε στόχους, αλλά μόνο στους ε, τομείς που αφορούν το ETS. Μόνο εκεί χρειαζόμαστε δεσμευτικούς ε, στόχους. Χρειαζόμαστε, όπως είπα, στόχους, προϋποθέσεις για το πώς αυτοί θα επιτευχθούν και, όπως υπόθηκε, χρειάζεται αυτή η δέσμευση να είναι παγκόσμια. Σωστά είπε και ο συνάδελφος Ρόιλ επίσης ότι υπάρχουν διαφορές από κράτος σε κράτος και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη και να το συνδυάσουμε με το παγκόσμιο γίγνεσθε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρίχαρτ Τζέμπερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την κοινή συζήτηση δύο επιτροπές. Ξέρω το άρθρο 51 δεν είναι ιδιαίτερα προσφυλέ στη διοίκηση του Κοινοβουλίου, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στη διαμόρφωση ε, των απόψεων και την αποκριστάλλωση εν ώψη ε, το ε, ε Χάρηκα πολύ που άκουσα Δανέζα Σοσιαλίστη να παραθέτει την Άγγελα Μέρκελ και η Γερμανία θέλει να έχει εθνικό στόχο 40% στο διοξίδιο του άνθρακα μείωση μέχρι το 2020, το μεγαλύτερο βιομηχανικό έθνος της Ευρώπης, μείων 40% μέχρι το 2020. Ακούω ότι και ο Κάμερον θέλει να το ρίξει στο μισό μέχρι το 2030 εάν υπάρξει και εφόσον μέχρι το 2015 διεθνή συμφωνία. Οπότε φαίνεται να κινούνται τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο. Ο δικός μας στόχος εδώ πρέπει να είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή λύση, να βρούμε μια τέτοια λύση και παραμένει η άποψή μου ότι τα δύο προβληματικά παιδεία, ενέργεια και προστασία του κλίματος είναι αλληλένδετα. Επίσης είναι μια κατάσταση εποφελής και για τα δύο μέρη, win-win. Οι τεχνολογίες που είναι φυτικές προς το κλίμα ε, δεν ε, είναι κατά της ευρωπαϊκής ανάπτυξης στην οικονομία. Γιατί ακριβώς αυτές οι τεχνολογίες που ε, πουλούν και πουλούνται αυτές που είναι στραμμένες προς το μέλλον. Και το δείχνουν και οι στατιστικές. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε διεθνώς την επαπαλαιωμένη τεχνολογία παρά μόνο τη σύγχρονη. Και εκεί θα πρέπει να επενδύουμε. Γι' αυτό είμαι πεπισμένος και εγώ ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτούς τους τρεις στόχους. Γιατί το είπε και ο Λάινεν αν διατηρήσουμε μόνο το στόχο του διοξιδίου του άνθρακα θα έχουμε μόνο πυρηνική ενέργεια και άνθρακα με CCS. Πώς θα γίνει όμως αυτό. Ε, τα κράτη με ελέγχουν τεράστιες διαφορές και έχουμε και μια κλασική αγορά. Η ενεργειακή ασφάλεια ε, δεν ε, μπορεί να υπολογιστεί σε κανένα τιμολόγιο. δεν υπολογίζεται η αξία της. Και ο στόχος του διοξιδίου του άνθρακα τελικά βρίσκει μεγάλη αντανάκλαση στις τιμές. Το ETS λέμε, υποτίθεται ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Κοιτάξτε τις στατιστικές. Η Δανία ε, πληρώνει 36 cents την κιλοβατόρα τον οικοκυριό Εμείς στην Αυστρία 20 cents. Ξέρετε ότι έχουμε και εκλογές το Σαββατοκυριακό. Το βιομηχανικό ρεύμα είναι 13 cents την κιλοβατόρα. Ποιο λέει ότι δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, να προσαρμόσουν τα εθνικά φορολογικά του συστήματα αν είναι πολύ ακριβό το ρεύμα. Και το βιομηχανικό ρεύμα δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην Ευρώπη από την Αμερική. Εντάξει, κάναν την επανάστασή τους στο λιθικό αέριο οι Αμερικανοί και έχουν τεράστια πλέον εκτήματα, αλλά οι τιμές ε, της ηλεκτρικής ενέργειας μόνο έμεσα συνδέονται με όλες αυτές τις ιστορίες. Παρακαλώ, ε, μην κάνουμε δογματικές και ιδεολογικές συζητήσεις, αλλά ρεαλιστικές. Να παραμείνουμε σε αυτούς τους τρεις στόχους. Ασφάλεια επενδύσεων να προσφέρουμε και αυτό είναι προς όφελος της οικονομίας και της βιομηχανίας και των θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ. Αυτή την προοδευτική ομιλία δεν ήθελα να τη σταματήσω καθόλου. Ε, από την Ήτρε, η συνάδελφος Ανδρέας Μπαρέα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, μια που βρίσκεται και στην καρδιά της ε, επίλυσης της κρίσης και είναι οικονομική λύση. Χρειαζόμαστε οικονομικές στρατηγικές, ε, μακροπρόθεσμα για την έρευνα, για την καινοτομία. Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα ήδη υπόθηκε είναι τεράστια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παράγουμε τίποτα απορρικτά. Γι' αυτό ε, είμαστε έρμεο των ε, εισαγωγικών. Το κανονιστικό πλαίσιο, ε, είπε ο Πρόεδρος, είναι κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ενιαία αγορά ενέργειας, να μεταφέρουν στην νομοθεσία του στα κράτη την ευρωπαϊκή υπόθεση. Ας πούμε, τα δίκτυα, η στενοποίη, αυτά τα bottlenecks, θα πρέπει να λυθούν τα ζητήματα. Έγινε λόγος ε, για το ότι δεν θα πρέπει να τα ποντάρουμε όλα σε ένα χαρτί, να έχουμε ένα και μόνο στόχο. Αυτό με τις ανανεώσιμες ήδη ισχύει στην Ευρώπη. Παράγουμε με διάφορους τρόπους, από το βορρά μέχρι το νότο της Ευρώπης. Υπάρχει, γίνεται αυτή η προσπάθεια και μπορούμε να παράγουμε ενέργεια χωρίς να χρειαζόμαστε εισαγωγές. Η βιομηχανία πρέπει να το λύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά και το θέμα της τιμής της ενέργειας, της πρόσβασης στην ενέργεια και να υπάρχει ένα κοινό κριτήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν πρόκειται να βρει λύση ούτε η βιομηχανία, ούτε η ίδια η κρίση σε τελική ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Χαίρομαι που βλέπω πολλούς συναδέλφους από την Επιτροπή Βιομηχανίας και πάλι, γιατί 7,5 χρόνια εργαζόμουν στην Επιτροπή αυτή και όταν το 2005 αρχίσαμε να συζητούμε για αυτούς τους στόχους, έτσι για πρώτη φορά. Και πολύ σημαντικό θεωρώ το γεγονό αυτό ότι συνεργαζόμαστε οι δύο επιτροπές. Ε, το κάνουμε έτσι και αλλιώς στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τώρα διακομματικά μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό και καλό είναι να είναι και διαφανές. Ποια είναι η αφετηρία μου εμένα για τη συζήτηση. Αυτό που είπε και ο Ρίχαρτ Ζέμπερ. Ότι το Ενωμένο Βασίλειο έκανε μια πρόταση η κυβέρνηση της αυτής μεγαλειότητος υπό την ηγεσία του David Cameron έχει καταθέσει επίσημα ένα έγγραφο που λέγει «Μέχρι το 2030 επιθυμούμε μείωση του διοξιδίου του άνθρακα στο μισό παρακαλώ». Και νομίζω ότι θα πρέπει από κοινού να το κοιτάξουμε αυτό, ιδιαίτερα... Παρακαλώ τον αγαπητό μου φίλο Κόνραντ Σιμάνσκι να το συνυπολογίσει, γιατί ο Ντέιβιτ Κάμερον είναι ο εφευρέτης και εμπνευστής της ομάδας ECR. Αν δεν τα είχε στυλώσει ο Κάμερον, δεν πρόκειται ποτέ να έχετε την ομάδα σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές. Αλλά και ο πολιτικός ρεαλισμός λέγει ότι το 50% αποκλείεται να έρθει. Είναι ενδιαφέρουσα μεν η πρόταση, πλην όμως ανέφικτη. Σίγουρα θα ε, υπολοιπόμεθα τα πολύ ε, το 2030. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου λέει και κάτι άλλο όμως ταυτόχρονα, ότι βάζουμε και όρους. Αν συμφωνήσει και το Παρίσι 40% ε, αλλιώς, μάλλον 50% αλλιώς 40%. Το είπα και στον Πολωνό Υπουργό προχτές. Σωστή είναι αυτή η μέθοδος. Ήδη με την Κοπεχάγη να βάγει σε αυτή η υπόθεση. Γιατί να λειτουργήσει τώρα στο Παρίσι. Μπορεί να έχουμε διαφορετικούς τρόπους και όλα ανεξάρτητα από τις ε, παγκόσμιες συμφωνίες, αλλά προτείνω να πούμε, ε, να κάνουμε αυτό που θεωρούμε μακροπρόθεσμα σημαντικό και σωστό. Και μετά το Παρίσι να συζητήσουμε. Θέλουμε να τελειώσουμε την κλιματική πολιτική, θέλουμε να την αποδυναμώσουμε, να πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Και τέλος, να υποστηρίξω πολύ αυτό που είπε ο Ζέμπερ, τρεις στόχους. Τα λέει και η συνθήκη αυτά έχουμε συμβατική υποχρέωση, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να τις ε, προωθούμε και όχι εις βάρος της ενεργειακής απόδοσης να τα υπολογίζει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ενεργειακή απόδοση, όχι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα και τις ανανεώσιμες, γιατί τότε μας συμφέρει και είναι και πιο φτηνό και αυτό θέλουμε όλοι. Ευχαριστώ, καλή πρόταση. Η κυβέρνηση Κάμερον. 50% αφού θα έχουμε και κυβέρνηση με τους πρασίνους δική σας στη Γερμανία, κάτι θα γίνει. Ο Κλώτ Τούρμας. I think that climate and... Νομίζω ότι το κλίμα και η ενεργειακή πολιτική πρέπει να είναι ένα ενιαίο πακέτο. Επειδή τρει στόχοι είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να δει κανεί τα πολιτικά πράγματα. Για δύο λόγου. Πρώτα απ' όλα, φανταστείτε πού θα βρισκόμασταν στην Ευρώπη εάν είχαμε μόνο το σύστημα ανταλλαγή ε, δικαιωμάτων εκπομπών έως σήμερα. Αυτή που λένε ότι το ETS ε, θα αρκούσε ή ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργούν ε, την, το πλώσμα στο ε, σύστημα, δεν είναι σωστό. 2,5 εκατομμύρια άδειες παραπάνω υπάρχουν και είναι περισσότερα αυτά ε, που αναγνωρίζουν στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Λιγότερα μάλλον από αυτά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, οι διεθνεί πιστώσει έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση το ETS και επειδή υπάρχει πάνω από ένα δι από παραθυράκια με 560 εκατομμύρια έλλειψη από, λόγω τη κρίση. Η τελευταία δεκαετία ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Εάν, και δεν θα έχει οδηγήσει πουθενά αν βασιζόταν μόνο στο ETS. Ο δεύτερο λόγο που οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και η πρέπει να προωθηθούν είναι ότι βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να περιορίσουν τη διακύμανση των τιμών και του κόστους και να είναι ένα ε, οικονομικό κίνητρο και μια οικονομική επένδυση. Έχει δίκιο ο Πίτερ Λίζε. Όσο καλύτερο modeling κάνει κανείς, όσο περισσότερα πρότυπα σχεδιάσει, τόσο περισσότερη αποδοτικότητα θα πετύχει. Περισσότερα μπορεί να πετύχει ως προς το στόχο του 50% λιγότερη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Ε, Αλλιώ με το ETS ε μπορεί να φτάσει στα 55-60 ευρώ τον τόνο για να το πετύχει. Εάν επιδιώξει κανείς 40% στόχο αποδοτικότητας, το 40% ανανεώσιμα και 50% αέρια του θερμοκηπίου μπορεί να πετύχει το 50% αέρια του θερμοκηπίου με 30 τιμή διοξείδιο του άνθρακα ανά τόνο. Διότι όλα τα μέτρα αποδοτικότητας που θα πυροδοτηθούν θα είναι φτηνότερα φτηνότερα γιατί θα είναι δεσμευτικά νέα σπί... Ε, καινούργια σπίτια, ε, στόχοι αποδοτικότητα, στόχοι για το διοξείδιο του άνθρακα, για τα ψυγεία, για το αέριο. Μπορούμε να πετύχουμε φτηνότερα μέτρα με δεσμευτικού ενεργειακού στόχου από ότι με την τιμολόγηση του διοξιδίου. Αυτοί λοιπόν που ανησυχούν για την οικονομία αυτή είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να πιέζουν ε, και να συνηγορούν υπέρ των στόχων αποδοτικότητας ως προς το θέμα των χωρών όπως η Πολωνία και άλλων. Να έχετε υπόψη το εξής και να μην ε, παραβλέπετε ότι η Πολωνία έχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό από ότι ε, να είναι ενεργειακά αυτάργης από ότι έχει δυναμικό σχιστολιθικό αέριο. Ε, το να μην υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι, τι σημαίνει δεν είμαστε πια αξιοπιστοί ως προς τα λόγια που λέμε για την ενεργειακή αυτάρκεια εάν τελικά δεν προωθούμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Χρειαζόμαστε στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί θα έχουμε αποτελέσματα. Θα έχουμε οικονομίες ως προς τα αέρια του θερμοκηπίου, στο χαμηλότερο κόστος και θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόληση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή ο Βιτόριο Πρόντι. Δύο λεπτά παρακαλώ. <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνεται να συζητήσουμε. Πρώτη παρατήρηση, το ETS δεν προχωρά. Νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να συζητήσουμε σε διαφορετική βάση. Στη βάση της κλιματικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, υλοποιώντας σε πολιτικό επίπεδο όσα διακηρύξαμε στο Μπαλί. Ακόμη και αν έχουμε διαφοροποιημένη προσέγγιση, αυτό που είχε χαρακτηριστεί ως differentiated responsibility. Ε, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το ETS, ας ξεχάσουμε και ας περάσουμε το φόρο για τον άνθρακα και να μην ξαναμιλήσουμε για το όλο θέμα. Επίσης, θα έπρεπε να καταργηθούν οι επιδοτήσεις των ορεικτών καυσίμων. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα και άλλο θέμα. Τέλος πάντων, θα πρέπει τώρα να κατανοήσουμε ότι οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις κλιματικές αλλαγές και το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, επιτόπου ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το έδαφος και να μπορέσει να προσαρμοστεί αυτό στις κλιματικές αλλαγές. Αυτή θα πρέπει να είναι η προϋπόθεση, η προϋπόθεση και η προτεραιότητα που θα πρέπει να μας καθοδηγήσει. Έπειτα υπάρχει το θέμα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μεταφορών. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ανανεώσιμες ενέργειες, ιδιαίτερα τον άνεμο, αλλά με ένα δίκτυο υψηλότατης ε, ε, αποτελεσματικότητας ως προς τη μεταφορά αυτής της ενέργειας. Θα πρέπει να βασιστούμε στο ανεξάντλητο δυναμικό του ανέμου. Αυτό ξεκαθαρι... δείχνει ξεκάθαρα μάλλον ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκών διαστάσεων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να επιληθεί. Δεν μπορούμε να το επιλύσουμε αμέσως, αλλά η εποδοτικότητα των ανανεώσιμων μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με ευρωπαϊκή παρέμβαση. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που μας απασχολεί, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς η ίδια η αλλαγή της νοοτροπίας θα δώσει ε, την ευκαιρία και στα άειλα αγαθά να ε, προστατεύονται και όχι μόνο στα υλικά τα οποία εκπροσωπεί το ΑΕΠ, θα πρέπει και αυτά να μετρώνται. Η Φιώνα Χολ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο σκιώδη συζητητή ε, τη ΑΛΔΑ για την Επιτροπή περιβάλλοντο, κύριο Γκεμπράντη, μου ζήτησε να διαβάσω τη δήλωση του εκ μέρου του. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή η κοινή συνεδρίαση και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με όλους εσάς έτσι ώστε να υλοποιήσουμε μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα για το 2020. Συζητώντας το πλαίσιο για το 2020, συνειδητοποιούμε ότι οι επενδύσεις ε, που κάνουμε τώρα θα έχουν επιπτώσεις ε, πολύ μετά το 2020 ε, το 2030 και χρειάζεται λοιπόν να το έχουμε αυτό υπόψη. Το, η διάσκεψη για το κλίμα των Ηνωμένων Εθνών το 2015 θα πρέπει να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει φιλόδοξους στόχους. Το πλαίσιο για το 2020 χρειάζεται να είναι φιλόδοξο για πολλούς λόγους. Καταρχάς πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους, τη μείωση ε, εκπομπών αρίων των θερμοκηπίου κατά 30% μέχρι το 2050. Αυτός όμως δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός μας ε, στόχος. Μια φιλόδοξη πολιτική θα πρέπει να στηρίζει την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να διασφαλίσει την, ε, τον ενεργειακό εφοδιασμό μας και να μας κάνει ενεργειακά αυτάρκης. Για να τα κάνουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε αποτελεσματικές πολιτικές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τρεις αποτυχίες του συστήματος της αγοράς. Ε, καταρχάς ε, την, σε αντιμετώπιση σε Τη μείωση των ε, εκπομπών αερίων μέσω χρήσης ανανεώσιμων ε, πηγών. Καταλαβαίνω ότι αυτή η στόχη είναι πολύ φιλόδοξη και φυσικά η τιμολόγηση του άνθρακα θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο για το πλαίσιο μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τώρα παρά αργότερα και να θέσουμε νέους στόχους για τους ε, τομείς ε, που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ωστόσο, δεν πρέπει να κοιτάξουμε εξετάζουμε μόνο την ετοιμολόγηση του άνθρακα, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα και η ενεργειακή κατανάλωση. Και αυτές οι επιδοτήσεις εκεί πρέπει να καταργηθούν, κατά την άποψή μου. Η τιμολόγηση του άνθρακα και μόνο δεν θα αρκέσει για να τονώσει τις επενδύσεις στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση. Χρειαζόμαστε και άλλους συμπληρωματικούς στόχους για το 2030 και οι στόχοι αυτοί θα συνεχίσουν να δίνουν την πολιτική όθηση μαζί με τα κριτήρια αξιολόγησης και με τους ε, πολιτικούς ε, στόχους. Ένα τέτοιο φιλόδοξο πλαίσιο θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να παραμείνει ε, πρωτοπόρος στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην τεχνολογία ανανεώσιμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή ο κύριος Αρσένης. Και δύο λεπτά. Α, απεχώρησε. Καλά. Μια σύντομη παρατήρηση τη κύρια Ουλσκοκ. Σύντομα είπαμε. Eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, να επιστρέψω σε αυτό που είπε ο κύριος Ρόιλ αν κατάλαβα καλά, είπε ότι υπάρχουν ορισμένοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα που είναι αντίθετοι σε ένα μείγμα ενεργειακό και υποστηρίζουν μόνο τις ανανεώσιμες. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα έχουμε ένα τέτοιο μείγμα χρήσης ενέργειας όπου οι ανανεώσιμες είναι ένα πολύ μικρό μέρος του. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για ένα μείγμα ως αποτέλεσμα. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις έτσι ώστε να προχωρήσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση προς μια, προς μια άλλη κατεύθυνση, προς μια αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που υπόθηκαν για τις επιδοτήσεις. Πολλοί από εσά θα αναφέρατε το θέμα αυτό εξάλλου, ότι είναι λάθος να στηρίζουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρησιμοποιώντας κρατική βοήθεια και κρατικές ενισχύσεις. Το γεγονός είναι ότι τώρα οι επιδοτήσεις είναι τεράστιες ε, στην πυρηνική ενέργεια και στην ε, ενέργεια από άνθρακα, ενώ οι επενδύσεις για τις ανανεώσιμες και επιδοτήσεις είναι πολύ χαμηλές. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για επενδύσεις στις ανανεώσιμες έχουν τεράστια προβλήματα. Δεν γνωρίζουν τις προϋποθέσεις που εμείς έχουμε θέσει για να είναι επιλέξιμοι για επιδοτήσεις και αυτό δεν οδηγεί σε μια ενεργειακή ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Η Γιολάντα Χούπνερ. Ευχαριστώ πολύ αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να συνδέσουμε την ενεργειακή και την κλιματική πολιτική, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, πώς θα επιδράσει αυτό και πώς θα την επηρεάσουμε άμεσα και ε, πώς αυτή θα επηρεάσει άμεσα την ε, εξέλιξη και την ίδια μας τη ζωή, ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργεί. Ε, κάτι που μου έρχεται στο μυαλό είναι η αστάθεια των κανόνων αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να αναλογιστούμε πώς το σύστημα θα γίνει πιο σταθερό. Έπειτα, πρέπει να αναλογιστούμε τις οικονομικές ε, συνέπειες αυτού αυτής της ε, ρύθμισης. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πράγματι είναι πολύ καλές πηγές ενέργειας, ωστόσο εξαρτάται από το πώς τις χρησιμοποιούμε. Δεν υπάρχει καμία μορφή τεχνολογίας που να ή που να μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε την ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίθετα υπάρχουν αντίστοιχες τεχνολογίες για, το, για την πυρηνική ενέργεια, για το φυσικό αέριο Χρησιμοποιούνται όμως πολύ λίγα χρήματα για επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια, για παράδειγμα. Μετά, χρειάζεται επενδύσεις, μεγαλύτερες επενδύσεις για τις νέες τεχνολογίες και δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για καλές ή κακές τεχνολογίες. Όχι. Μιλούμε για πηγές ενέργειας, δεν μιλάμε όμως για την ουσία. Η ουσία είναι οι νέες μέθοδοι, οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Πρέπει να μπορέσουμε να δείξουμε στη νέα γενιά έναν ορίζοντα και γι' αυτό χρειαζόμαστε επενδύσεις και έτσι θα λύσουμε πολλά προβλήματα. Ο Γιώλα Λάινεν θα ήθελε να κάνει μια σύντομη παρατήρηση. Ναι. Ακριβώς αυτό που είπε η Γιολάντα Χίπνερ πρέπει να συμβεί μέχρι το 2030. Πρέπει αυτό το σύστημα να συμπληρωθεί, να ολοκληρωθεί, διότι έχει ελλείψεις. Λείπουν τα έξυπνα δίκτυα, τα smart grids, λείπουν οι αποθηκευτικές δυνατότητες, λείπουν οι νέες τεχνολογίες στην αγορά, χρειαζόμαστε όθηση, χρειαζόμαστε κίνητρα για επενδύσεις και χρειαζόμαστε και δυνατότητα και αγορά δυνατοτήτων. Είναι σίγουρα κάτι που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε backup όταν θα κλείσουμε τα εργοστάσια, ε, τα συμβατικά εργοστάσια. Διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα. Και εδώ πρέπει να επενδύσουμε. Να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επενδύσουν και τα κράτη-μέλη. Ε, τώρα, όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχω να πω ότι η τιμή Τις ενέργειες από ανανεώσιμες πηγές έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες τώρα δείχνουν ότι η ολική ενέργεια είναι ανταγωνιστική. Στην, ε, ιδιαίτερα στην κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας. Το ίδιο και για το βιοαέριο και ε, υπάρχουν βελτιώσει από πλευράς ε, ποιότητα Και α μην κοιτάμε στο παρελθόν. Εντάξει, στο παρελθόν ήταν πιο, ακριβά, ε, πιο ακριβές οι τιμές και η Γερμανία σε αυτόν τον τομέα στι ανανεώσιμε ήταν όντως πρωτοπόρος. Χρησιμοποίησαμε φωτοβολταϊκά. Όμως έγιναν τόσο μεγάλες επενδύσεις που στον που μειώθηκε η τιμή. Και θα σταματήσω εδώ γιατί μίλησα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε δύο εκπρόσωπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο από του δύο θα ήθελε να μιλήσει. Εσεί, ε, γάμα δέλτα κλίμα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ήσασταν και χθε εδώ όλοι, ο πρόεδρο. Είναι μια κοινή επιτροπή, γι' αυτό είμαι και πάλι εδώ. Η ΓΔ Κλίμα συνεργάζεται πάρα πολύ και με τι δύο επιτροπέ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην συναδελφό μου κυρία Κρίστοφερ λίγο μετά να πω ότι η συζήτηση αυτή μέχρι τώρα ήταν αρκετά πλούσια. Όπω ξέρετε, ο πρόεδρος Σαμπαρόζο στην ομιλία του για την κατάσταση τη Ένωση, παρουσίασε ορισμένε προτάσει, είπε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένε προτάσει μέχρι το τέλο του χρόνου και συνεργαζόμαστε και με τι άλλε υπηρεσίε τη Κομισιόν για το θέμα αυτό. Και το Μάρτιο του 2004 θα έχουμε νεότερα. Φυσικά καλωσορίζουμε τις προσπάθειες που κάνετε, τη δουλειά που κάνετε και την ε, συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη των στόχων του 2030. Δύο λόγια γιατί τώρα κάνουμε αυτές τις ενέργειες. Δύο είναι οι λόγοι, δύο είναι τα ζητήματα και πολλοί από σας είπατε πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Βασικά από, το πλευρά, από τη μεριά του κλίματος Έχουμε την εδέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, η μελέτη και η έκθεση για αυτή θα δημοσιευθεί αύριο και σε σχέση επίσης και με τις ε, επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Και με, με λίγα λόγια να σας πω ότι όλες οι χώρες ε, συμφωνούν προς ε, μία κοινή λύση, ότι πρέπει να βρεθεί μια κοινή λύση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ενωμένη εν ώψη της, διάσκεψης, ε, της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα, να μιλήσει με μία φωνή και έχουμε μία ευκαιρία. Διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα και όχι μόνο αυτές και η Κίνα και από την Κίνα βλέπουμε πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίε που έχουν αναλυφθεί και για τι ανανεώσιμε και για πιλωτικά ε, προγράμματα ETS. Υπάρχει λοιπόν ευκαιρία εδώ να προχωρήσουμε τους στόχους και χρειαζόμαστε αυτή την παγκόσμια συμφωνία για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό και πρέπει να μιλήσουμε με μια φωνή. Επίσης, όσον αφορά την ενέργεια, πάρα πολλοί από εσά αναφέρατε την εξάρτηση που έχουμε από τις εισαγωγές την αύξηση στις τιμές των καυσίμων και η κατάσταση στην Ευρώπη έχει ως εξής. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πλέον τα προβλήματά μας, τα οποία και όλα έχουν και είναι και συνδεδεμένα με το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Και σε αυτό στοχεύει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα δημοσιευτεί. Επίσης, έχουμε, απαντήσει, έχουμε λάβει πολλές απαντήσεις από διάφορους ενδιαφερόμενους πάνω από 500 απαντήσεις νομίζω από διάφορους εφορείς και μαζί με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από το πακέτο θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε μια περιεκτική πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που μόλις ε, ακούσαμε. Για μας είναι σημαντικό, ακούστηκε άλλωστε, να έχουμε τρεις στόχους ανταγωνιστικότητα, αηφορία και δυνατότητα εφοδιασμού σε ενέργεια για το 2030. Τώρα εργαζόμαστε για μια μελέτη αντικτύπου που επίκειται αρχές Οκτωβρίου θα δρομολογηθεί για να έχουμε μία βάση, να μπορέσουμε να εργαστούμε με σενάρια και να προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε διάφορα μοντέλα και διάφορους στόχους για να έχουμε και κάποιες ενδείξεις για το τι μέλη γενέστε και ποια πορεία μπορούμε να ακολουθήσουμε. Διδαχτήκαμε από το πακέτο για το 2020, μπορούμε να σας συμπεριλάβουμε εκεί. Κάναμε και διαβούλευση και συζήτηση με τα κράτη-μέλη και ένα τύπο συμβούλιο ενέργειας, αλλά και η συζήτηση δεν σταματά εδώ. Θα, ε, πρέπει να σας πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας και στο μέλλον, αλλά η σημερινή συζήτηση μας ικανοποίησε πολύ. Ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο στους δύο συνεισηγητές, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, πολύ σύντομα. Ναι, ζήτησα το λόγο γιατί μίλησαν και άλλοι περισσότερες φορές. Και λέω, αφού μπορούν αυτοί, μπορώ κι εγώ, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν έπρεπε. Είναι προνόμιο για ορισμένους. Για σας πάντα. Ναι, γι' αυτό ξαναζήτησα το λόγο. Μπορώ. Ωραία. Έχω μια επικριτική παρατήρηση σε δύο σημεία. Άκουσα ότι ορισμένοι συνάδελφοι διαφώνησαν με τον ένα στόχο, γιατί ένας στόχος σημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί και από την πυρηνική ενέργεια ε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Μα αυτό είναι έολο το επιχείρημα ποιο ενεργειακό μείγμα επιλέγουμε και ποια ενεργειακή ε, πολιτική, αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Αν έχουμε εμεί τρεις στόχους ή κατά ενός στόχου, έχοντας στο μυαλό μας τι θα υπαγορεύσουμε και τι θα απαγορεύσουμε στα κράτη-μέλη, ε, καλή επιτυχία. Κάποιοι συνάδελφοι είπανε ότι και βέβαια οι ανανεώσιμες πηγές έχουν ε, επιπτώσεις ε, στα πιστοποιητικά, στο, στην τιμή και τα λοιπά. Ενδιαφέρον είναι αυτό, άρα υπάρχουν επιδράσεις, ανεπιθύμητες παρενέργειες, άρα δικαιούται κανείς να αναρωτηθεί. Ο πρώτος στόχος, πώς επιδρά στο στόχο νούμερο 2 ή στο στόχο νούμερο 3. Και μήπως θα ήταν καλύτερο να υπάρχει μια ιεράρχηση αυτών των στόχων σας το δίνω αυτό προσκέψη αν ζητάτε να σκεφτούμε για αυτά τα θέματα ακόμα. Μα τι είναι αυτό. Μα γι' αυτό δεν ήρθαμε εδώ, έχετε αμφιβολίες, ακριβώ για να σκεφτόμαστε, για να ανταλλάσσουμε απόψεις και ο Κλωτούρμος που θέλει και αυτός να τα ξαναπεί. Ωραία, αρχίσαμε δεύτερο γύρο. Χέρμπερτ, είπες ότι αλληλεπιδρούν οι ανανεώσιμες με το κλίμα. Για θυμίσου λίγο τους αριθμούς που έδωσα. 2,2 δισεκατομμύρια ε, από το ETS. 50 εκατομμύρια τα οφείλουν στις ανανεώσιμες. Γιατί δεν είναι παραπάνω. Γιατί ήδη από το 2006 όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε το πακέτο της για το 2020, γιατί ήδη από τότε συμπεριέλαμβανε στους υπολογισμούς τις ανανεώσιμες. Σήμερα τι βλάπτει το ETS, όχι οι ανανεώσιμες. Ακούς, Χέρμπερτ. Ένα παραθυράκι που το 2004 τελευταία ώρα έβαλε η Business Europe, International Credits. Λέγαμε καλά δεν πειράζει, βάλτε το γι' αυτό. Ναι, αλλά τώρα καταλάβαμε ότι αυτό σημαίνει 1,1 δισεκατομμύρια ε, περίσευμα μισό σέντ έκανε ε, το 2011 ο τόνος για να το αγοράσουν και επίτηδες ε, να βάγισε το σύστημα γιατί το τορπίλησαν. Και όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα με το ETS, αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα, τις διεθνείς πιστώσεις, το International Credits και επίσης πώς θα δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο με το, μεταξύ του στόχου ε, ETS ε και της ανάπτυξης της οικονομίας. Και έχω και μια ερώτηση, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει ο κύριος Βεργό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, η Κομισιόν υπολογίζει μέχρι το 2030 η οικονομία να αυξάνεται ετησίως με ρυθμούς της τάξης του 1,4% ή 1,8%. Υπάρχει κανένας εδώ μέσα που να πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία την επόμενη 20 ετία 17 εν πάση περιπτώσει χρόνια θα αυξηθεί κατά 1,4 και 1,8%. Δηλαδή το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να κάνει μια ανάλυση ευαισθησίας. Δηλαδή αν είναι αυτό 1% πώς μετακυλείεται μετά ο υπολογισμός. Εμείς πώς μπορούμε να κάνουμε εδώ πολιτική εάν τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιείται δεν συνάδουν αν μη τι άλλο με την πραγματικότητα. Κανένας δεν γνωρίζει πώς και αν θα επιβεβαιωθεί αυτό. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε δύο υπολογισμούς, μεγάλη ανάπτυξη και μικρή. Και το 50% αέρια του θερμοκηπίου με πιθανή ε, μεγέθηση της οικονομίας που δεν θα φτάνει στο 2%, τι θα σημάνει και, τι, ε, και πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή οικονομία να το επιμειστεί, γιατί θα έχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και πολύ περισσότερες ανανεώσιμες. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα δύο συναδέλφους, κυρίες, η κυρία Γιόρνταν Σίσελ και η Σάτου Χάση και θα ήθελα να κλείσω τον κατάλογο. Εκτός αν ανοίξουμε πάλι τον κατάλογο από τα, πίσω προς τα εμπρός, γιατί έχουμε χρόνο, να μην ξανακάνουμε συζητήσεις. Θέλει κανένας άλλος το λόγο. Όχι. Ωραία, κλείνει εδώ ο κατάλογος και μετά οι συγητές. Η Ρωμάνα Γιόρνταν. Komentirati želim predvsem eh, to, da so mnogi kolegi... Ναι, να σχολιάσω μόνο κάτι. Πάρα πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για σταθερότητα και ότι πρέπει να στοχεύσουμε στην σταθερότητα. Όλοι θέλουμε τη σταθερότητα, αλλά υπάρχουν δύο βασικές διαφορετικές προσεγγίσεις. Οι μεν θέλουν επιδοτήσεις, οι δε θέλουν να σταματήσουν οι επιδοτήσεις. Μετά, η άλλη προσέγγιση είναι περισσότερο οικονομική. Ο κύριος στόχος μας είναι φυσικά η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και πρέπει για να γίνει αυτό να λάβουμε υπόψη και την αγορά. Η αγορά είναι κάτι δυναμικό, κάτι που εξελίσσεται το οποίο όμως μπορούμε να σταθεροποιήσουμε με πολιτική θέληση. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα, αλλά αυτό δεν θα γίνει αν η πολιτική κάθε χρόνο αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αναφέρθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο ως παράδειγμα, με τους υψηλού στόχους της μείωσης εκπομπών. Κανείς όμως δεν είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει τεχνολογικά ουδέτερο. Έχουν έναν στόχο και τα υπόλοιπα θα τα αφήσουν στην αγορά. Η αγορά θα ρυθμίσει τα πάντα. Θα ρυθμίσει λοιπόν το ποιες τεχνολογίες θα αναπτυχθούν περισσότερο. Κλοντ, συμφωνώ μαζί σου με το ETS και με τα προβλήματα που προκαλεί. Προβλήματα όμως δεν προκαλεί μόνο το ETS, προβλήματα προκαλεί και η τιμή του άνθρακα. Και αυτό προκαλεί και το πρόβλημα της δυσκολίας στην πρόσβαση στην αγορά, στις νέες τεχνολογίες. Και τώρα κάτι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσατε για μία ανάλυση. Εμένα θα με ενδιέφερε σε αυτήν την ανάλυση αν ε, ε, υπάρχει και συμπεριλαμβάνεται ένα σενάριο με όλους και τους τρεις στόχους μαζί της ε, μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ε, κυρία Σατουχάση, ευχαριστώ πρόεδρε. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα πρέπει στο μέσο ενός αγώνα να αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Όταν λοιπόν συζητούμε τους κανόνες για το 2030, πρέπει να είμαστε σαφείς ότι θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα που να λειτουργήσει εύρυθμα, που να είναι, να είναι ε, σε θέση να λειτουργήσει. Δεν πρέπει να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια. Οι επιστήμονες λένε ότι οι κλιματικές αλλαγές πρέπει να αντιμετωπιστούν κατεπηγόντως. Και όλες οι σχετικές μελέτες λένε ότι όσο νωρίτερα αναλάβουμε δράση για να τις αναχαιτήσουμε, τόσο περισσότερο θα εξοικονομήσουμε ως προς το κόστος. Όσο καθυστερούμε την ε, δράση, τόσο μεγαλύτερο κόστος θα πρέπει να καταβάλουμε. Ε, απλώς λοιπόν ε, είναι σαφές ότι οι λόγοι είναι οικονομικοί για να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Φέτος, πριν από λίγους μήνες, η Ολλανδική Υπηρεσία Περιβαλλοντικών ε, ε, Συλλογήσεων είπε ότι κατά 80-90% επιτεύχθηκαν δεν θα επιτευχθούν μάλλον οι στόχοι περιορισμού των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε κατά ένα 80% ε, με μόνο δράση για το διοξίδιο του άνθρακα. Όχι. Πρέπει να στηρίξουμε τους στόχους της ενεργικής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ίδιο είπε και ο Παγκόσμιο Οργανισμό περιβάλλοντος ότι δεν φτάνει ο μετριασμός εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Χρειάζονται και οι υπόλοιποι στόχοι. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι όσοι είναι ε, σοβαροί και το εννοούν αυτό για τους μακροπρόθεσμους στόχους, το καταλαβαίνουν. Χρειαζόμαστε και συμπληρωματικούς κι άλλους στόχους. Τους ε, στόχους της ανανεώσιμης ενέργειας, την αποδοτικότητα της ενέργειας. Αυτή και πιο σταθερή είναι και πιο μόνιμη και λιγότερο διακειμένοντας προς τις τιμές. Δεν είναι όπως η εμπορία ε, των δικαιωμάτων εκπομπών. Οι ανανεώσιμε πηγέ, η ενεργειακή αποδοτικότητα ε, επιτρέπουν μεγαλύτερη βεβαιότητα και ασφάλεια για τι επενδύσει. Ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλο. Κυρία Χούμπνερ, μόλι έκλεισα το κατάλογο των ομιλητών. Δεν μπορώ να σα βάλω. Καλά. Ε, εντάξει. Συγγνώμη. Αλλά η συνάδελφος απευθύνεται σε μένα. Να απαντήσω λοιπόν, θέλω μόνο. Δεν μπορεί να αλλάζει διάδρομο ένα άλογο στον υπόδρομο την ώρα του αγώνα. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε ούτε να αλλάζουμε κι εμείς άλογος καβαλάριδες την ώρα του, της κούρσας. Οι κανόνες για το μέλλον πρέπει να είναι σαφείς, πρέπει να γίνουν τώρα όμως, πρέπει τώρα να γίνει ο σχεδιασμός τους. Τώρα πρέπει να καθορίσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, ακόμα τις απόψεις όλων αυτών των οργανισμών, του επιχειρηματικού κόσμου, αυτούς που είναι υπέρ, αυτούς που είναι κατά, αυτούς που αγοράζουν την ενέργεια. Λοιπόν, αυτά πρέπει να γίνουν τώρα και όχι στο μέλλον. Λοιπόν, ωραία. Και ερχόμαστε τώρα στους δύο συν ο Κόρατσι πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε όλους όσοι έκαναν να παρατηρήσεις εδώ, αλλά δεν είναι δυνατό. Θα σταθώ λοιπόν σε ένα-δυο σημεία μόνο, που τα επανέλαβαν οι περισσότεροι συνάδελφοι. Κατά πρώτον, η ευθύνη μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ Είμαι ένας νέος βουλευτής και ακούω με ιδιαίτερη προσήλωση και προσοχή τις απόψεις των συναδέλφων. Τα όσα λέει ο, ο ΙΕ. Εδώ θα υπάρξει επιστημονική αξιολόγηση για το τι συμβαίνει με το κλίμα. Όμως δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το κόστος ε, των κλιματικών αλλαγών σωστά μετράται. Εάν δεν έσφαλα τα τελευταία χρόνια ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίων, ο υπόλοιπος κόσμος έχει περιοριστεί σε δηλώσεις, σε λόγια τα οποία ακούσαμε πρόσφατα και από τον πρόεδρο Ομπάμα. Δεν συμφωνώ λοιπόν με τον μεγάλο μας ενθουσιασμό. Πρόκειται για μια πολιτική στρατηγική. Βλέπω εδώ να υπάρχει μια τάση να καθησυχάζονται οι πολιτικές ανησυχίες των διαφορών χωρών. Όμως τα γεγονότα λένε κάτι διαφορετικό. Ζούμε σε μια περίοδο και ζούμε μια στιγμή όπου πρέπει να κινητοποιηθούμε. Χρειαζόμαστε αέριο. Είμαστε εκτεθειμένοι στις ανάγκες μας αέρια και χρειαζόμαστε φθηνό αέριο στην Ευρώπη. Αυτό είναι κατά πρώτον πολιτική ευθύνη. Δεν είναι προβλητική η ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολλές οι οικονομίες που μπορούν ε, να αναπτυχθούν ακολουθώντας το δικό μας το παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μας ως υπόδειγμα. Αυτές τις πολιτικές επιλογές πρέπει να κάνουμε, ώστε αυτές οι οικονομίες να ε, στριμωχτούν, να τις κολλήσουμε στον τοίχο διότι δεν μπορούν να αρνηθούν τα χειροπιαστά γεγονότα. Δεύτερο σημείο, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Είναι μια πολύ σημαντική πηγή αυτή για να αντλήσουμε ενέργεια στο μέλλον. Όχι μόνο από περιβαλλοντική σκοπιά, αλλά και γιατί οι ενεργειακοί μας πόροι μπορούν να τονώσουν την ενεργειακή αγορά, να εξασφαλίσουν την τροφοδότηση και την προμηθεία μας ενέργεια εδώ πρέπει να ακολουθήσουμε όμως και το ρυθμό των εξελίξεων. Και υπάρχει ε, ένα μεγάλο πεδίο για να συζητήσουμε εδώ. Είναι πολύ ευρύ το θέμα. Συζητούμε για επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές και το κατά πόσον θα είναι κερδοφόρες. Η πολιτική. η Πολωνοί, η πράσινοι Πολωνοί έκρωσαν τον κόδωνα του κινδύνου για τη χρήση της βιομάζας σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά δεν είναι άστοχα στο συγκεκριμένο θέμα και στη συγκεκριμένη συζήτηση. Έχουμε πολύ ψηλέ προσδοκίε σε όλα τα κάτι μέλη και ταυτόχρονα πολλού ενδιασμού για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο στόχος λοιπόν αυτός ε, πρέπει να γίνει μια πεποίθηση για όλη την Ευρώπη. Γιατί για την ώρα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από χώρα σε χώρα. Και έπειτα το θέμα είναι τι γίνεται και με την αξιολόγηση. Γιατί έχουμε μια τεράστια δυνατότητα να ε, υπάρξουν εδώ συνέπειες. Είναι μεγάλη σφαίρα της επιρροής μας το πώς θα ε, κατευθύνονται τα κονδύλια για το κάθε ε, μέτρο, για την κάθε μας πολιτική, είναι πολύ σημαντικό. Η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα λόγω χάρη είναι κάτι που πραγματικά είναι δαπανηρό. Πρέπει να σκεφτούμε αν αυτό θα ωφελήσει, αν θα έχει θετικό αντίκτυπο στις μεταφορές. Ο άνεμος μπορεί να μην είναι αποτελεσματική πηγή ενέργεια στη στιγμή που υπάρχουν, που υπάρχουν ατανάξει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ε, πρημοδοτούν λόγω χάρη τι ανανεώσιμε πηγέ για να αντιμετωπίσουν τι κλιματικέ αλλαγέ. Η αποτέφρωση του άνθρακα και η έκκληση των αερίων στην ατμόσφαιρα είναι κάτι που οι Ηνωμένε Πολιτείε το συνεχίζουν. Οι εκπομπέ λοιπόν των αερίων του θερμοκηπίου είναι αυτέ που πρέπει να έχουμε υπόψη μα. Όχι μόνο δείκτε δείκτες που να είναι χαρακτηριστικοί. Όταν λοιπόν συζητούμε τέτοια θέματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα θέματα αυτά είναι σοβαρά για το μέλλον. Σήμερα έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πεποίθηση. Το κόστο ε, ε, του περιορισμού εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα δεν μπορεί να μας κάνει να παραβλέπουμε την οικονομική κρίση. Υπάρχει επιβράδυνση στην οικονομική ανάπτυξη. Τα κόστη και το κόστος γενικά θα είναι υψηλό, αλλά μπορεί να περιοριστεί εφόσον κάνουμε περισσότερες επενδύσεις. Υπάρχει ασύμμετρη λοιπόν ανάπτυξη στα διάφορα μέτρα που θα επιλέξουμε ενδεχομένω και κυρίως από οικονομική σκοπιά στο μέλλον. Θέλουμε ο να φτάσει στην τιμή των 30 ευρώ μέχρι το 2030. Όμως πρέπει στις Βρυξέλλες να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας και να αναλάβουμε να αποφασίσουμε τα σωστά μέτρα. Το οφείλουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν έχουν να κάνουν με τις ανανεώσιμες πηγές ή όχι. Ούτε με, την, με το επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχουν να κάνουν με την εναρμόνιση των στόχων. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να διαθέτουν και ευελιξία. Είναι πολύ διαφορετική η στάση των ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ του και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια νέα προσέγγιση. Ευχαριστώ. Η Άντελ τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω καταρχά να ευχαριστήσω όλου όσοι ε, συνεισέφεραν και εμπλούτησαν πολύ τη συζήτηση. Ε, και θέλω να επιμείνω, δεν θα πρέπει η θεώρηση να είναι περιοριστική. Είναι πάρα πολλέ οι ε, υποθέσεις που διακυβεύονται εδώ. Να μην το περιορίζουμε. Εγώ θα εξακολουθήσω να ζητώ ένα πακέτο, μία δέσμη με τρεις στόχους. Μου φαίνεται εκ των όνων κάνευ. Να συνεχίσουμε σε αυτή την ατραπό, σε αυτή την κατεύθυνση και να δούμε επιτέλους ποιες είναι οι συνέπειες ενεργείες μεταξύ των τριών πόλων που μας απασχολούν τόση ώρα. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτή η προσπάθεια, εκεί θα πρέπει να εργαστούμε. Στη συνδυασμένη πρόοδο χρειάζεται πολύ περισσότερη βελξία. Και ξέρετε τι με κάνει έτσι λίγο να γελάω σήμερα. Στη συζήτηση για την ε, εμπορία εκπομπών και το backloading είναι... δείχνει ότι οι ίδιοι μας λέγουν ότι σήμερα θέλουμε να έχουμε ένα πακέτο με ένα στόχο που να βασίζεται σε ένα ε, ισχυρό ETS. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ξαφνικά αλλάζουν γνώμη. Και πολύ. Και θυμίζω τους εν λόγω ότι χωρίς ε, ενεργειακή απόδοση και χωρίς ανανεώσιμες η τιμή του διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να είναι πολύ πιο υψηλή και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας έγινε λόγος για επιδοτήσεις. Συμφωνώ απολύτως και θα πρέπει και αυτό να το ξεκαθαρίζουμε. Υπάρχουν επικαλύψεις οι οποίες είναι απαράδεκτες μεταξύ των ε, εθνικών ενισχύσεων και των ευρωπαϊκών. Σας μίλησα για σταδιακή εγκατάλειψη, ένα είδος phasing out, γιατί έχω συναντηθεί με τον κλάδο των ανανεώσιμων. Οι ίδιοι μας το πρότειναν ότι είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί πλέον και γίνεται αυτή ε, η δυνατότητα. Ε, είναι δυνατό. Και εμείς ε, έχουμε ε, την αιωλική ενέργεια. Στη χώρα μου έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας, τις χερσές ανεμογεννήτριες. Τώρα θα πρέπει να πάμε στο πέλαγος. Ένα τρίτο ενδιαφέρον να πούμε στον κύριο Σιμάνσκι ενδεχομένως. Θέλω και εγώ να θυμίσουμε τη σημασία της έρευνας, της ανάπτυξης και και να πούμε ότι θα πρέπει να παραμένουμε ανταγωνιστικοί παγκοσμίω. Δεν μας περιμένουν οι άλλοι. Μιλήστε για την Κίνα. Τον Ιούλιο η Κίνα ανακοίνωσε 200 δισεκατομμύρια δολάρια στις ανανεώσιμες επενδύσεις. Το καλοκαίρι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα κύριε Σιμάνσκι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν στόχους μείωσης ε, ε, εκπομπών ε, αερίου συγγνώμη, θερμοκηπίου. Βέβαια το συζητούν ακόμα γιατί δεν συμφωνεί το Κογκρέσο, αλλά ο, ο πρόεδρος Ομπάμα το έχει διατρανώσει αυτό ως βούληση. Επίσης έγινε λόγους για την αξιοπιστία. Ναι, πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι για να έχουμε και πρόσωπο διεθνώς. Δεν μπορούμε τη μια μέρα λέμε άσπρο και μετά από λίγες μέρες μαύρο. Για μένα η συνέπεια ε, και η συνέχεια έχουν σημασία. Και η αξιοπιστία ε, είναι να μιλάς με μία φωνή εξ ονόματος της Ευρώπη και όχι εξ ονόματος της χώρας του ο καθένας, εξ ονόματος της Ευρώπης και θέλω να το τονίσω αυτό. Γίνεται λόγος για επιμερισμό ε, της προσπάθειας. Effort sharing. Ναι, και η Πολωνία και η Γαλλία και άλλες χώρες να έχουν συλλογική συζήτηση. Και όχι χώρα με τη χώρα. Και ε, τέλος, όταν μιλώ για αξιοπιστία, δεν ήμουν εδώ στο Κοινοβούλιο όταν αποφασίστηκε η δέσμη για το κλίμα. Ήμουν εκτός, ήμουν στη, στη Βελγική Γερουσία και χαιρόμουν πάρα πολύ για τη φιλοδοξία που έβλεπα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα, βέβαια πέρασε και η κρίση έκτοτε και το ξέρω ότι είναι προτεραιότητα, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι το κλίμα δεν είναι πια επίγον. Και ορισμένοι που ήταν παρόντες ε, τότε και συμμετείχαν, ε, σήμερα έχουν αλλάξει τακτική και στάση, λες και έχει εξαφανιστεί η κλιματική αλλαγή. Μα εμείς έχουμε ευθύνη ως νομοθέτες να κοιτάμε όλες τις τυχές οικονομικές, κοινωνικές, κλιματικές ε, και άλλες και όχι να εθελοτυφλούμε λέγοντας ότι άλλαξαν οι προτεραιότητες, γιατί παραμένει επίγουσα η κατάσταση και για την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω ε, αν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε. Τελειώσαμε. Η κυρία Σαρτόρη έχει το λόγο, η πρόεδρος της Επιτροπής ε, Βιομηχανία. Παρακαλώ. Προσωπικά και απλώς ε, σε προσωπικό επίπεδο να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρότε για τη δουλειά του, για το συντονισμό των εισηγητών ε, και της συζήτησης ήταν πλούσια συζήτηση και πολύ χρήσιμη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές διαφορετικές απόψεις, είναι πολλοί οι τομείς που εμπλέκονται εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι ο διάλογος μεταξύ των ε, συναδέλφων από το Κοινοβούλιο και των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, της ΕΝΒΕ και της ΙΤΡΕ, θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε ξεκάθαρες διότι εάν δεν είμαστε αρκετά ε, έτοιμοι για να συμφωνήσουμε, διευκρινήσεις και περαιτέρω εξηγήσεις μπορεί να υπάρξουν μεταξύ μας, δεν είναι θέμα αυτό. Θα ξαναβρεθούμε εδώ στις 7 Νοεμβρίου, θα συνεννοηθώ με τον συνάδελφο Γκρότε, νομίζω ότι και πάλι θα τα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία να έχουμε ταυτόχρονη συνεδρία, κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρτόρη. Ε, να ευχαριστήσω ξανά τη γραμματεία, τους συναδέλφους. Μπορούμε να συνηθίσουμε έτσι ωραία αυτό το άρθρο 51, να το κάνουμε πιο συχνά. Μπράβο, μπράβο στη γραμματεία και μπράβο σε όλους. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε ευθύνη, επαναλαμβάνω, καταρχάς ως θεσμικό όργανο και φοβάμαι ότι χωρίς μια ξεκάθαρη θέση θα υποχωρήσουμε, θα πάμε πίσω σε μια επανακρατικοποίηση της ενεργειακής πολιτικής και της κλιματικής πολιτικής. Πρέπει να μιλήσουμε και για το δίκαιο του ανταγωνισμού Πρέπει να μιλήσουμε για τα εθνικά συσχήματα ενισχύσεων και πώς αυτά θα λειτουργήσουν στο μέλλον. Τι χρειάζεται η βιομηχανία. Χρειάζεται ρεύμα. Αλλά και αυτό χρειάζεται ρυθμίσεις. Δεν μπορούν οι τιμές του ηλεκτρισμού να αυξάνονται συνέχεια και χωρίς τέλος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η κυρία Χιούπνερ το είπε, δεν πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Εδώ έχουμε επίσης να πω και έναν νέο, τη μελλοντική γενιά, έναν νέο της μελλοντική γενιάς των φιλελεύθερων, ενδεχομένων, ο οποίος μόνο να κερδίσει θα έχει από την πολιτική που πρέπει να κάνουμε. Και να κάνω μια έκκληση σε όλους ξανά. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, ένβη ή ήτρε. Κύριε Σιμάνσκι, όλοι προερχόμαστε από διαφορετικά κράτη-μέλη και πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να μην κοιτάζει ο καθένας το συμφέρον του. Πρέπει να βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες του καθενός, να τις λαμβάνουμε υπόψη και έτσι να πορευόμαστε και να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα αντανακλά τις θέσεις όλων. Στις 17 Νοεμβρίου η κυρία Σαρτόρη θα προεδρεύσει τη συνεδρίαση. 12 Νοεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Στις 2 Δεκεμβρίου θα συζητήσουμε στις τροπο, ε, τροπολογίες και θα ψηφίσουμε από κοινού στις 9 Ιανουαρίου του 2014. Ελπίζω και οι συγητές και οι σκιώδες συγητές να είναι υπεύθυνοι και να συνεργαστούν καλά. Εντάξει, μπορούμε όλοι να έχουμε τις διαφωνίες μας, όμως έχουμε μια κοινή ευθύνη. Ξανά, 3 μέχρι 6 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε. και ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά. Να ευχαριστήσω ξανά τους εισηγητές, τους και εισηγητές και όλους όσους βρέθηκαν εδώ. Ευχαριστώ πολύ.